I think we can start. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ενδεχομένω. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εκπληκτικό ότι ενώ είμαστε τόσο κοντά στα Χριστούγεννα, βρίσκονται τόσοι πολλοί από εμά στην αίθουσα. Έχουμε λοιπόν τις τελευταίες συνδυάσει μας εφέτος. Ξεκινώ με την έγκριση τη προσωρινή ημερησία διάταξη εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσει. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχουν, αλλά θα ήθελα εγώ να σα πω το εξή για τους ε, Ο κύριο Σασόλη θα έλθει ε, να μας πει για τα θέματα της διακυβέρνηση και για τον τρίλογο για τα τεχνικά θέματα θα έχουμε μια παρουσίαση για τα θέματα αυτά σε λίγο. Πρακτικά της 3ης Δεκεμβρίου, εάν δεν υπάρξει αντίληση, θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί. Ερχόμαστε τώρα στην παρουσίαση της GDMU για την έκθεση της Κομισιόν για τις κοινέ προδιαγραφές και τα πρότυπα για τους οργανισμούς ε, ελέγχου των πλοίων και τους οργανισμούς υποπτίας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καραμήτρο. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά περίπου. Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, good afternoon to all of you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους σας. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αναφερθώ κυρίως στο άρθρο 10 που κατά τη γνώμη του κυρίου Τεγκράντες που ήταν και ο πρωτεργάτης αυτού του θέματος ε, δεν είναι εδώ σήμερα αλλά το γνωρίζει πολύ καλά. Καταρχήν να σας ε, πω περί τίνος πρόκειται. Τι είναι αυτές οι επιθεωρήσεις, οι επιθεωρήσεις των πλοίων. Γίνονται από τις ε, εταιρείε ταξινόμησης, τους νεογνώμονες. 50 είναι ανά τον κόσμο και 11 χρησιμοποιούμε νεογνώμονες εμείς για τα δικά μας σκάφη. Αναγνωρισμένες δηλαδή ε, από, τα, την Ευρωπαϊκή Ένωση οργανώσεις, ε, οργανισμούς μάλλον. Τα κράτη σημαίες μπορούν να, ε, να δώσουν σε αυτούς τους οργανισμούς την δυνατότητα να κάνουν επιθεωρήσεις και να δώσουν πιστοποιητικό. Μάλιστα είναι θέματα καταστατικής επιθεώρησης, καταστατικού ελέγχου για θέματα που προβλέπουν και υποχρεώνουν οι διεθνείς συμβάσεις τα κράτη σημαίας να ζητήσουν αναγνώριση. Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιτρέψουν σε εταιρείε πιστοποίηση μόνο εφόσον αυτέ είναι αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, τέτοιοι, τέτοιοι νεογνώμονες έχουν κανόνες και τεχνικά πρότυπα που είναι ιδιωτικά και που χρησιμοποιούνται από τους νεογνώμονε για να εξακριβώσουν και να ε, πιστοποιήσουν ότι ακόμη και η κατασκευή, η ολόκληρη κατασκευή του πλοίου συνάδει με τις προδιαγραφές. Έχουμε δηλαδή αφενός τις νόμιμες ε, υποχρεώσεις από τις διεθνείς συμβάσεις και έχουμε και τις ιδιωτικές υποχρεώσεις από τους αναγνωρισμένους τους οργανισμούς. Το αποτέλεσμα αυτού του έργου πιστοποίησης είναι ότι οι νεογνώμονες δίνουν ένα πιστοποιητικό κλάσης. Αυτό το πιστοποιητικό ε, διευκολύνει τον πλειοκτήτη να συνάψει ασφάλιση. Και από τη στιγμή που γίνεται η πιστοποίηση θεωρείται ότι έχει το πιστοποιητικό κλάσης και άρα μπορεί να πλέψει. Αυτά ως προς τεχνικές προδιαγραφές ε, για την αναγνώριση των πιστοποιητικών ε, κλάσης. Επίσης είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία πιστοποίησης λαμβάνει υπόψη όλα τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πλοίου. Καθένα από αυτά έχει και ατομικό πιστοποιητικό. Και όλα ε, πιστοποιούνται από την ε, εταιρεία αυτή της αναγνώρισης, αυτόν τον αναγνωρισμένο οργανισμό. Αυτό αναφέρονται στον κανονισμό που προβλέπει αμοιβαία αναγνώριση. Η αυτό προβλέπει ότι οι εταιρείε πιστοποίηση ε, αναγνωρίζουν αμοιβαία τα πιστοποιητικά του, ώστε ο κατασκευαστή να μην χρειάζεται κάθε φορά ο πλειοκτήτη ε, να πηγαίνει και να ζητάει από κάθε εταιρεία το πιστοποιητικό. Γιατί τη μία φορά προτιμώ τη μία ε, εταιρεία πιστοποίηση και την άλλη φορά την άλλη. Θέλουμε λοιπόν για να μειώσουμε το κόστος μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση και να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών αυτών των ε, εταιριών, των υιογνωμόνων. Είχαμε μακρά συζήτηση και με τη βιομηχανία και τον κλάδο και νομίζω ότι είναι προς όφελος και των δύο πλευρών αυτή η συμφωνία, η ρύθμιση. Και για τον κλάδο γιατί κάθε φορά που παρασκευάζεται ένα προϊόν δεν θα πρέπει να πηγαίνει ε, σε κάθε ξεχωριστή εταιρεία πιστοποίηση που θέλει να χρησιμοποιήσει ο πλειοκτήτης και ο ίδιος εξοπλισμός για το ίδιο εργαστήριο και για τον ίδιο σκοπό πολλές φορές πιστοποιείται διαφορετικά με πλέον κόστος κάθε φορά και επίσης και για τους νεογνώμονες ε, χάνεται χρόνος ε, και χρήμα. Ενώ αν έχουμε αμοιβαία αναγνώριση και εναρμόνιση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και στις υψηλότερες προδιαγραφές, αυτό ωφελεί και την ασφάλεια αλλά και την φήμη αυτής της ε, εταιρείας πιστοποίησης. Φαίνεται αυτό εύκολο ίσως στη θεωρία, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο στην πράξη. Γιατί, όπως σας είπα, οι εταιρείε πιστοποίηση έχουν τους δικούς τους ιδιωτικούς κανόνες, που μερικές φορές διαφέρουν κιόλα μεταξύ τους. Οπότε, στο δικό μας ε, ε, κανονισμό προβλέπεται ότι τα, οι πιο απαιτητικέ και αυστηρές προδιαγραφές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από όλε τι εταιρείε πιστοποίηση. Έχουμε 11 τέτοιε εταιρείε, ε, του νεογνώμονε δηλαδή. Θα πρέπει να καθίσουν και να συμφωνήσουν ποιε είναι οι αυστηρότερε προδιαγραφέ και αυτέ να ισχύουν για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί η πιστοποίηση δίνεται για πολλά και διάφορα θέματα. Αυτό είναι καλό για τη βιομηχανία, γιατί ο κλάδος απασχολεί περίπου 450.000 ε, εργαζομένους με πλήρη απασχόληση. Και επίσης ε, για τους προμηθευτές ο τζίρος είναι 125 δισεκατομμύρια περίπου και μάλιστα το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 43%. Οπότε αν ο κατασκευαστής ε, κάθε φορά και για κάθε δομικό στοιχείο, για κάθε πλοίο πρέπει να ζητά διαφορετική πιστοποίηση εξαιτία ε, των πολλών νεογνωμόνων που είναι από πίσω, το κόστος είναι υπέρογο κάτι που πλήττει την ανταγωνιστικότητά του απέναντι στους ιδούς Κινέζους ε, ή άλλους κατασκευαστές είναι και προς το βιομηχανικό συμφέρον, δηλαδή προς το συμφέρον της βιομηχανίας να προωθήσουμε αυτή την εναρμόνιση. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να τονίσω εδώ είναι ότι αυτή η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών κλάσης στηρίζεται στον κανονισμό ε, για την ασφάλεια και την εταιρική σχέση με τη βιομηχανία. Γιατί Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αναγνωρισμένων Εταιριών και είναι η ομάδα της αμοιβαίας αναγνώρισης που συστήθηκε από τις ίδιους τους νεογνώμονες καταρχήν για να διαχειριστούν τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων που εμπίπτουν στον καθεστώς της αμοιβαίας αναγνώρισης, να βρουν τους τρόπους και μεθοδολογία μεταξύ τους, ε, να παράσχουν και ένα συγκεντρώνουν τη τεχνογνωσία που χρειάζεται, να εντοπίσουν τα προϊόντα που εμπίπτουν σε αυτό το καθεστώ αμοιβαία αναγνώριση, γιατί δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια και έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά πολλέ φορέ. Και βέβαια να τεκμηριώσουν και να σχεδιάσουν κριτήρια αξιολόγηση και τεχνικέ προποθέσει. Μάλιστα, αυτή η ομάδα καθόρισε ότι τα προϊόντα που εμπίπτουν στην αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία έγκριση τύπου. Μέχρι στιγμή έχουν 44 ομάδες το τελευταίο 1,5 χρόνο μετά από συνεννοήσεις κατέληξαν σε 44 τέτοια προϊόντα που εμπίπτουν στο καθεστώ τη αμοιβαία αναγνώριση. Ποιο είναι το πλεονέκτημα. Εκτό ότι μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων πιστοποιητικών, είναι, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των κατασκευαστών, γιατί περιορίζει τη γραφειοκρατία. Επίση, οι κατασκευαστέ ε, έχουν πρόσβαση σε μια παγκόσμια αγορά πολύ πιο ευέλικτη γιατί δεν χρειάζεται κάθε φορά για κάθε δομικό στοιχείο, για κάθε προϊόν να ζητούν ξεχωριστό πιστοποιητικό. Τώρα, και κάποια άλλα σημεία που αναφέρονται. Μια και είναι σχετικά καινούργιο αυτό το σύστημα και είναι και εθελοντικό. Είναι δηλαδή μια βιομηχανική διαδικασία που πρέπει να γίνει σεβαστή και μέχρι στιγμή λειτουργεί. Προϋποθέτει την ανάμειξη των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα αυτό ισχύει για τους μικρομεσαίους κατασκευαστές που δεν γνωρίζουν όλες τις δυνατότητες και που δεν είναι εξοικειωμένοι, δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτού του καθεστώτος αμοιβαίας αναγνώρισης. Ένα άλλο θέμα που ίσως ε, έχετε λάβει υπόψη είναι ότι η διεθνής αναγνώριση του καθεστώτος αυτού δεν είναι προφανής. Γιατί κάποιες, ε, κάποια κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατασκευαστές που δεν είναι Ευρωπαίοι ίσως κρίνουν ότι αυτό το σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης παρεμποδίζει τη δική τους πλήρη ελευθερία. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι γενικώ η εφαρμογή του καθεστώτος αυτού συνάδει και με τον κανονισμό. Βέβαια έχουμε ακόμη μερικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, το σύστημα αυτό, το καθεστώς αυτό ε, στηρίζεται στην αρχή της αυτορύθμισης και της εταιρική σχέσης με τον κλάδο. Αυτή η εταιρική σχέση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του καθεστώτος για την οργάνωση, την εφαρμογή και την τακτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. Η εμπειρία είναι πολύ σημαντική και θα είναι σημαντική και για το μέλλον. Και είναι φυσικό ότι θα πρέπει να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Όπως σας είπα, είναι θέμα αυτορύθμισης και κάτι τέτοιο πολλές φορές είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ε, ακριβώς επειδή είναι εκούσιο θέμα. Πάντως, δεδομένης έκδοση των νέων πιστοποιητικών, μπορούμε να έχουμε θετικά στοιχεία και ικανοποίηση. Και επειδή υιοθετούνται τα αυστηρότερα πρότυπα και προδιαγραφές, νομίζω ότι είναι προς όφελος και του κατασκευαστών και των πλειοκτητών που έχουν μικρότερο γραφειοκρατικό κόστος, αλλά υπέρ και της ασφάλειας των πλοίων, γιατί είναι αυστηρότερες προδιαγραφές που ισχύουν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι χάρη στην πρωτοβουλία αυτή έχουμε ένα επιπλέον στοιχείο που προσθέθηκε στον κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτερ Φαντάλεν, ναι. Ποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Δύο, τρεις, τρεις ομιλητές. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι πρωτού γίνω μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εγώ είχα ασχοληθεί με τα θέματα αυτά στις ε, κάτω χώρες. Είναι πολύ καλό να αναγνωρίζετε όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά τι γίνεται με την... Ε, τι γίνεται με την εποπτεία αυτών των ε, εταιριών, των νεογνωμόνων. Όταν ήμουν εγώ λοιπόν διευθυντής του φορέα επιθεώρησης της κάτω χώρες, είχα διαπιστώσει ότι υπάρχουν φυσικά διαφορές μεταξύ των ιογρομόνων και οι φορείς αυτοί οι οποίοι δίνουν πιστοποιητικά ως νεογρόμονες στην Ευρώπη δεν είναι συγκρίσιμοι με τους αντίστοιχους οργανισμούς στην Ασία. Παρά το γεγονός ότι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Πώς λοιπόν μπορούμε να εξασφαλίσουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή διαδικασία έγκρισης για ευρωπαϊκούς νεογνώμονες και με ποιο τρόπο η Κομισιόν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές μεταξύ παραγωγή των γραφείων μια, ενός νεογνώμονα στην Ευρώπη και στην Ασία. Και αυτό έχει να κάνει με τις διαφορές στην αυπηγική ε, διαδικασία που ακολουθείται εκεί. Ευχαριστώ κύριο Κάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Καραμίτσος έχει ήδη αναφερθεί στο όνομα του Λούις Τεγράνδες, ο οποίος φυσικά είναι στη Μαδρίτη, όπως μπορείτε να φανταστείτε, <clears throat> γιατί συνεχίζεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πρόσφατων εκλογών στην Ισπανία. Και φυσικά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ ζωντανή μέρα αυτή στη Μαδρίτη. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Καρανίτσο για τις πληροφορίε που μα έχει δώσει. Αλλά έχω κάποια ερωτήματα για τη λειτουργία του άρθρου, για τη χρήση του άρθρου 10. Από ό,τι έχω ακούσει. Ο ιδιωτικό τομέα, ο οποίο ουσιαστικά ε, είναι ένα είδος οργανισμού ομπρέλας σε σχέση με τους νεογνώμονες, λειτουργεί με μεγάλη βραδίτιδα. Αυτό όμως έχει σημαντικές ε, επιπτώσεις στη λειτουργία των νεογνωμόνων, γιατί οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να προβαίνουν σε κάποιες αξιολογήσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολυδάπανες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα αυτό, ιδίω για την αυπηγική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνονται γρήγορα οι αξιολογήσεις αυτές. <clears throat> Κύριε Καραμίτσο λοιπόν, έχετε ε, μία εξέταση για τα διάφορα επίπεδα από το επίπεδο 1 έως το επίπεδο 6. Εσείς ελέγχετε όλους τους τομείς αυτούς ή τους ουσιαστικά επιφορτίζετε τα, τους νιογνώμονες με τον έλεγχο αυτών των ε, επίπεδων. Επίσης η ομάδα μας θα ήθελε να ξέρει καλύτερα και για το χρονοδιάγραμμα το οποίο αφορά τις αμοιβέ αναγνωρίσεις. αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στον κανονισμό και αυτό μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του κανονισμού στην περίπτωση που, παραδείγματος σε πέντε χρόνια, θα είναι δυνατόν να σταματήσει η προκατακτική διαδικασία για την αμοιβαία αναγνώριση και γίνει πραγματικότητα η αμοιβαία αναγνώριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζω ότι έχετε μεγάλη εμπειρία για το πακέτο <clears throat> για τα ναυτικά θέματα που περάσαμε πριν από 10 χρόνια και ξέρουμε πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία αρμόσει και ζήνε μάλιστα τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καρανίσο και πάλι που είναι μαζί μας για την έκθεση που μας έχει δώσει. Είναι πάρα πολύ καλό να, αυτά που, να ακούσουμε αυτά που είπε. <clears throat> Εγώ έχω μόνο ένα ερώτημα. Είπατε ότι η διεθνής αναγνώριση είναι ένα δύσκολο θέμα. Και φυσικά είπατε ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι γίνεται με τους δικούς μας νεογνώμονες και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους νεογνώμονες της Απανατολής Παγκοσχάρης, της Κίνας. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε υπό το πνεύμα της φιλελευθεροποίησης. Είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε ένα πιο γρήγορο βήμα στην αγορά με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Κούν. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, λέει ο κύριο Κούν, και εγώ φυσικά θέλω να εξασφαλίσω ότι θα υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν η εναρμόνιση των ε, ε διαδικασιών αξιολόγησης της κατασκευής των πλοίων. <clears throat> Πρέπει να γνωρίζει κανείς όταν φτιάνεται ένα πλοίο ποια υλικά χρησιμοποιεί, ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιεί, ποιες ε, ε δυνατότητες μηχανημάτων δίνεται σε ένα πλοίο, ποια είναι τα κινητήρια συστήματα, τα μηχανικά ενός πλοίου. Αν εγώ θέλω να δώσω παραγγελία για ένα νέο πλοίο, θα πρέπει να είναι σύμμορφα αυτά τα οποία προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός ε, Ναυτιλίας, ο IMO, και η Σύμβαση Όλας για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. Και μόνο τότε θα πρέπει να δημιουργούνται, να χτίζονται αυτά τα πλοία. Ακούσαμε ότι 43% των, ε, της προσθέμενης αξίας στην αυτοίγική και αυτό περιλαμβάνει και τους εργαζόμενους στην αυτοίγική βρίσκονται στην Ευρώπη. Αλλά είμαστε σε κάπως οριακή θέση στην αυτοιγεία σε ό,τι αφορά τα πλοία για κοντέινερ, τα πλοία για χίδιν φορτίο κτλ. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την, ε, τον ανταγωνισμό από την απαρατολή. Η Κορέα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και έχει κάνει πάρα πολλού αγώνες. Έχουμε κάνει πολλούς αγώνες για να αντιμετωπίσουμε την, ε, τις επιδοτήσεις που δίνονται στην αφήγικη βιομηχανία. Και το ερώτημα είναι, μπορούν οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές, και είναι πολλοί αυτοί από την Ελλάδα ω τη Γερμανία, ω άλλε χώρε τη Ευρώπη, μπορούν να εξασφαλίσουν οι εφοπλιστέ ότι όταν δίνουν μια ε, εντολή βάση αυτών που έχει αποφασίσει ένας νεογνώμονας θα τηρηθούν αυτές οι προδιαγραφές πλήρως στην Ευρώπη όταν μιλάμε εδώ για τους κινητήρες ή τις ε, έλικες των πλοίων που προερχόνται από το Μέκλεμπορκ παραδείγματος χάρη που μπορεί να πουλάνε έλικες ε, πρόθεση στην Κορέα ή στην Κίνα κτλ. μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνεται ο έλεγχος και η επαλήθευση για τον εξοπλισμό αυτό όπως γίνεται και στην Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί πια <clears throat> δεν είναι τόσο δυνατοί στα φορτηγά πλοία, κάνουν ε, κρουασιερόπλοια και άλλα επιβατικά πλοία. Αλλά αυτή τη στιγμή η κρουασιέρα, τα κρουαζιερόπλια βρίσκονται περισσότερο σε ευρωπαϊκά χέρια. Είναι απαραίτητο λοιπόν να τηρηθούν οι προδιαγραφές που θέλουμε εμείς και μας ενδιαφέρει να υπάρξει η σωστή προ... και επιστοποίηση όλων των στοιχείων ενός πλοίου, κυρίως των μηχανών που δίνουμε στα πλοία της Αποανατολής. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Κούν, ο οποίος είναι φανερό ότι είναι ναυπηγός και τα γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα αυτά. Ε, ε, Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε τεχνικά ζητήματα γιατί δυστυχώς δεν είμαι ναυπηγός, αλλά νομικός. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για αυτό το μηχανισμό που είναι πολύ σημαντικός. Συμφωνώ ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καλό θα ήταν να έχουμε αφενός αυστηρές προδιαγραφές, αφετέρου σαφείς προδιαγραφές ε, και πρότυπα για την κατασκευή και την ε, εκμετάλλευση του σκάφους. Βέβαια, ο μηχανισμός έγκυται στο ότι οι μονομένε χώρες ε, αναγνωρίζουν ότι τα σκάφη πληρούν τους συγκεκριμένους κανόνες. Τώρα όμως έχουμε την εξής κατάσταση. Δηλαδή, όταν η πιστοποίηση γίνεται από όργανα, από αρχές πολλών χωρών, από οργανισμούς πολλών χωρών, που οι πρακτικές τους μπορεί να διαφέρουν. Ερωτώ λοιπόν, προβλέπετε σε τέτοιες περιπτώσεις ένας ελεγκτικός μηχανισμός, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό αν μια χώρα είναι πιο επίοικης για παράδειγμα, πιο ανεκτική, έχουμε ένα ελεκτικό μηχανισμό για να επιθεωρήσουμε την κατάσταση, τις πρακτικές που ισχύουν ε, για, για ώστε να μην έχουμε διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω και πάλι στον κύριο Καρανίσο στην Κομισιόν το λόγο για να απαντήσει τις πολυπληθείς ερωτήσεις που τέθηκαν. Παρακαλώ. Thank you very much and Σα ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλε. τι ερωτήσει, αλλά συγχωρέστε με αν τυχόν κάτι μου διαφύγει. Να ξεκινήσω καταρχά. εξηγώντα το ζήτημα που αφορά το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο επίπεδο, το διεθνέ επίπεδο, διότι είναι σαφέ νομίζω πω ένα πλοίο το οποίο ταξιδεύει παντού θα πρέπει να ε, τηρεί τις ίδιες προδιαγραφές με τα υπόλοιπα που κάνουν την ίδια δουλειά. Δηλαδή ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκριση ε, για το κατά πόσο δηλαδή κάποιος εξοπλισμός ε, απευθύνεται σε ένα πλοίο που πλέει στα ευρωπαϊκά ύδατα ή στα διεθνή ύδατα. Θέλουμε να είναι όλα τα ίδια. Θέλουμε οι γνώμονες να ακολουθούν τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές. Αυτοί που είναι οι ευρωπαϊκοί, οι νιογνώμονες, το δέχονται σχετικά εύκολα, ενώ για να σας το πω ξεκάθαρα έχουμε αντιρρήσεις από εκείνους τους νεογνώμονες που βρίσκονται εκτός της ευρωπαϊκής ε, επικράτειας και που είναι αναγνωρισμένοι. Δηλαδή, ABS, που ήταν ε, ο ηγέτης ε, στη φάση της, ε, της αντιπαράθεσης, αμερικανικός νιογνώμονας, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς. Το ίδιο ισχύει και για τους κινέζικους, ιαπωνικούς ή κορεατικούς νιογνώμονες, διότι φυσικά αν, αν έχουμε αυτή την αμοιβή αναγνώριση χάνουν δουλειά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μεγάλος πόλεμος λοιπόν έγινε αλλά τουλάχιστον καταφέραμε να επιβάλλουμε την άποψή μας. Έχουμε διμερείς ε, βέβαια συμφωνίες με κάποιες άλλες σημαίες που λέμε ε, αυτό είναι το πρότυπο, είναι ψηλότερο από το δικό σας, ακολουθήστε το. Για να ξεκαθαρίσουμε, υπάρχει Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας, υπάρχουν δηλαδή οι προδιαγραφές καταστατικές ε, του, αυτού του Διεθνούς Οργανισμού και μετά είναι και η ιδιωτική. Δηλαδή ένα σκάφος αναγνωρίζεται, επειδή ίσως να τηρεί τα στάνταρ του ΑΕΜΟ, αλλά η ναυπηγική του, για να πούμε, ή ο αρχιτέκτονάς του, έχει ακολουθήσει την καλύτερη δυνατή προσέγγιση. Αυτά μπορώ να σας πω όσον αφορά τα ιδιωτικά πρότυπα αναγνώρισης, ιδιωτικού νεογνώμονες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι με αυτή τη συμφωνία τουλάχιστον ε, επειδή αυτές οι μη, ευρωπαϊκές, οι μη ευρωπαϊκοί νεογνώμονες συνεργάζονται μαζί μας για να εναρμονίσουμε τα χαρακτηριστικά και τα πρότυπα για ζητήματα όπως κάποια εξαρτήματα των μηχανών ή κάποια τμήματα των εξοπλισμών, τουλάχιστον εκεί χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια, τα ίδια στάνταρ για τη δική τους πιστοποίηση και δεν θα ζητήσουν από τον πλειοκτήτη να πληρώσει επιπλέον χρήματα για να πιστοποιήσουν ακόμα μια φορά έναν εξοπλισμό που έχει ήδη πιστοποιηθεί. Για τον ίδιο ιδιοκτήτη που έχει ένα άλλο καράβι με ευρωπαϊκή σημαία ή κινέζικη σημαία, αμερικανική σημαία. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά για να σας πω ε, ποιο είναι το συμφέρον των δικών μας κατασκευαστών καταρχήν να αποφύγουν τη διπλή ε, πιστοποίηση του ίδιου εξοπλισμού και απ' την άλλη να καταλάβουμε το συμφέρον των ιδιωτικών νεογνωμόνων που κάθε φορά θέλουν να μπορούν να πιστοποιούν το ίδιο, τον ίδιο εξοπλισμό εφόσον έχει κατασκευαστεί σε ένα άλλο ε, εργοστάσιο και έχει πιστοποιηθεί αλλού. Και για να απαντήσω και στον κύριο Κάμπα να πω ότι δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε όλους τους εξοπλισμούς. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε 43 ομάδες εξοπλισμών που είναι σχετικά πλούστεροι και που πλέον έχουν εναρμονιστεί ανάμεσα στους διάφορους νεογνώμονες. Και επίσης ε, τοποθετούνται σε σκάφη συγκεκριμένων κλάσεων σε κάθε εταιρεία, αλλά είναι κάτι που θα πάρει καιρό. Πάρα πολύ καιρό πήρε το να ξεκινήσει η διαδικασία. Το τελευταίο 1,5 χρόνο με χαρά είδαμε ότι επιταχύνθηκε η διαδικασία και ότι ο κόσμος συνεργάζεται περισσότερο και με μεγαλύτερη σοβαρότητα από ό,τι παλιότερα. Βεβαίως, εδώ η τα ευρωπαϊκά τμήματα μια εταιρεία ή τα ασιατικά τμήματα μια εταιρεία δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους εξοπλισμούς τους ή τα εξαρτήματα ανάλογα με το αν θα εγκατασταθούν σε ευρωπαϊκό ή κινέζικο πλοίο. Αυτό το επιληθεύουμε ούτως ή άλλως, να μην υπάρχουν διαφορές. Άλλα ερωτήματα. Κύριε Κούνε, μιλάμε για το 43% των κατασκευαστών εξοπλισμών. <clears throat> Όχι δυστυχώς για τα ίδια τα σκάφη. Δυστυχώς η μεγαλύτερη αξία ενό σκάφου δεν είναι ο εξοπλισμός, αλλά το ίδιο το χτίσιμο του πλοίου που αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο βαθμό γίνεται στην Ασία. Πάντως οι κατασκευαστές εξοπλισμών είναι σε το μεγαλύτερο αριθμό Ευρωπαίοι. 43% σας είπα των εξοπλισμών των σκαφών, των πλοίων θα ωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα διότι έτσι μειώνεται το κόστος τους μέσω τη της μείωσης των διοικητικών ε, ε, διαδικασιών. Στο τελευταίο τμήμα ίσω είναι λίγο πιο δύσκολο να το κατανοήσει κανεί. Πάντω, δεν είναι τα κράτη και οι αρχέ που αναγνωρίζουν όλα τα πρότυπα. Τα κράτη και οι αρχέ αναγνωρίζουν τμήμα των προτύπων που είναι τα χαρακτηριστικά του ΆΕΜΟ, τα πρότυπα του, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλία δηλαδή, που είναι τα στάνταρ των διεθνών συμβάσεων. Όλα τα υπόλοιπα που είναι η μεγαλύτερη αξία ω ποσοστό του σκάφου είναι τα πρότυπα των ιογνωμόνων που είναι όπω είπα ιδιωτικέ εταιρείε. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και το κόστος για τους ε, κατασκευαστές. Δεν ξέρω αν έγινα σαφής και αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Τουλάχιστον προσπάθησα να απαντήσω στα περισσότερα ερωτήματα. Αν έχετε κι άλλα βεβαίως θα μπορέσω ίσως στο τέλος της συνεδρίασης να κάνω κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις αν τα επιθυμείτε. Ευχαριστώ κύριε Φάντε Δύο ερωτήσεις θέλω, θέλω να επανέστω. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά, τελικά μπορούμε να βρεθούμε όμοιροι των ε, μη ευρωπαϊκών υιογνωμόνων. Αν βραδιπορούν αυτοί οι νεογνώμονες, τότε είμαστε δεμένοι χεροπόδαρα με αυτούς. <clears throat> Και το επόμενο ερώτημα είναι πότε μπορεί ο κύριος Καραμίτσος να μας πει ότι θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Αν έχει να μας πει κάτι για το χρονοδιάγραμμα. Γεια, yeah, Παρακαλώ, κύριε Καραμίτσο. Well, I'm not a... Δεν είμαι προφήτης. Ε. Δεν είναι δυνατό να ξέρει κανείς, γιατί πάντα έρχονται νέοι είδη εξοπλισμού για τα πλοία στην αγορά κτλ. Το γεγονό ότι εμεί προσπαθούμε να καταλήξουμε τουλάχιστον σε κοινού κανόνε για τα απλούστερα είδη ε, εξοπλισμού και να τα χρησιμοποιούν όλοι στο πιο ψηλό δυνατό επίπεδο, αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν για ιδιαίτερα είδη πλοίων εξειδικευμένοι εξοπλισμοί που δεν μπορούν να τύχουν εναρμόνιση μεταξύ νεογνωμόνων. Δεν θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Και υπάρχουν επίση εξοπλισμοί για ένα συγκεκριμένο είδο κινητήρο. Ούτε και αυτοί μπορούν να ε, μπορέσουν να εναρμονιστούν. <coughs> Έχουμε αυτή τη στιγμή 43 ομάδε εξοπλισμού στις οποίε εργαζόμαστε. Μπορεί να είναι μετά 100, μπορεί να είναι 120. Εμεί κάνουμε αυτή τη ε, διαδικασία με τη βοήθεια των τεχνικών ε, συνεργατών μας από τη Λισαβόνα, αλλά όλα αυτά θα απαιτήσουν μεγαλύτερη καλή θέληση θα έλεγα από την πλευρά των ιογνωμόνων για να προχωρήσουμε και φυσικά και κάποια μεγαλύτερη πίεση από τους κατασκευαστές εξοπλισμού, ιδίως από τις μεγαλύτερες τέτοιε εταιρείε που θέλουν διαδικασία πιστοποίησης να μην είναι τόσο πολύ δάπανη. Είναι μια διαδικασία που δεν θα τελειώσει αύριο, θα συνεχίσει και δεν μπορώ να σας δώσω κάποια ημερομηνία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι μια ατέρμονη διαδικασία. Νομίζω ότι ήδη αν μπορέσουμε 20-30% των εξοπλισμών να είναι αμοιβαία γνωρίσουμε, αυτό είναι ήδη μια μεγάλη ε, <clears throat> Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο επόμενο ε, στοιχείο της ημερήσια διάταξης So, wir kommen jetzt zur Präsentation des Ερχόμαστε στην παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικών για τα αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της συνδεδομικής υποδομής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που υπάρχουν οι εκπρόσωποι του Fraunhofer Institute, του M5, που είναι παρόντες. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο στον καθένα για πέντε λεπτά και μετά μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια να παρουσιάσετε τη μελέτη αυτή, η οποία έχει γίνει μετά από αίτηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προεπολογισμού, αλλά είναι προφανές ότι και εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών ενδιαφερόμαστε τα μάλα για το θέμα αυτό και σας δίνω λοιπόν το λόγο κύριε Σάντε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερω που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε την παρουσίαση αυτή τη συνεδρίασή σα. Ερχόμαστε εδώ, δεν είναι η πρώτη φορά. Είμαστε πάλι γνώριμοι και θα σα παρουσιάσω ευχαρίστω αυτή τη μελέτη για την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης ιδεροδρομικών υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είμαστε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, υποφαινόμενο ο Βέρνερ Ρόδενγκάτερ και ο Κλάους Ντόλ. Εμείς είμαστε οι βασικοί συντάκτες ε, της έκθεσης αυτής ε, του Fraunhofer ISI από τη Γερμανία. Για να δούμε αν μπορούμε να λειτουργήσουμε εδώ το μηχάνημα για τις διαφάνειες. Παρά είμαι γρήγορος για το σύστημα, δεν με προλαβαίνει. Καταρχήν να σας ενημερώσω για τους στόχους. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της μελέτης. Κυρίως ε, να απαντήσω στο ερώτημα πόσο αποτελεσματική είναι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των σιδηροδρόμων και αν ε, υλοποιεί τους βασικούς στόχους της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των κρατών μελών και της εύρυθμης λειτουργίας ε, της εσωτερικής αγοράς. Βέβαια και άλλα ερωτήματα τέθηκαν στη μελέτη μας. Για παράδειγμα, ποιος είναι ο αντίκτυπος των διαφόρων σιδηροδρομικών σχεδίων, ε, των προηγούμενων και των μελλοντικών και θέματα πολιτικής επίσης πολύ σημαντικά. Για το πώς να αναζωογονήσουμε τους σιδηροδρόμους, πώς να επιλέξουμε τα προγράμματα που έχουν την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συστηθέμενη αξία και ούτω καθεξής. Τέτοιου είδους ερωτήματα μας προβλημάτισαν κατά την εκπόνηση της μελέτης μας. Στην δεύτερη διαφάνεια ε, έχουμε ένα συνοθήλευμα αναλύσεων και συμπερασμάτων Καταρχήν, ποιοι είναι οι παράγοντε τη επιτυχία, ποιε είναι οι προποθέσει για μια επιτυχή πολιτική. Είναι ένα συνδυασμό βιβλιογραφία, έρευνα και συμπερασμάτων στα οποία καταλήξαμε μετά τι αναλύσει μα. Αν θέλουμε μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πολιτική για του σιδεροδρόμου και ένα ευρωπαϊκό σύστημα, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αισθενιστούν αυτή την προσέγγιση και από τεχνολογική πλευρά και από οργανωτική πλευρά στόχος φυσικά είναι να αναπτύξουμε, και αυτό οφείλουμε να κάνουμε, ένα ανταγωνιστικό σιδηροδρομικό σύστημα που θα είναι ανταγωνιστικό και στις μεγάλες αποστάσεις. Για τις άλλες χώρες όπως στη Βόρεια Αμερική, εκεί έχουμε πολύ επιτυχημένο σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλων αποστάσεων. Για να επιτύχουμε αυτή την ανταγωνιστικότητα λοιπόν, θα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως συνδεδεμένα σιδηροδρομικά δίκτυα, να εξαλείψουμε τις στενοπούς και τις συμφορήσεις και να εξυγχρονίσουμε το σιδηροδρομικό μας δίκτυο που δεν θα πρέπει να κολλάει σε... στις από τα σύνορα. Επίσης θα πρέπει να έχουμε πλήρως συνδεδεμένα δίκτυα με την κατάλληλη τεχνολογία και τα, σύστημα ελέγχου, ε, τα συστήματα ελέγχου επίσης να είναι διαλειτουργικά για να μην χρειάζεται να αλλάζουμε ε, τις ε, μηχανές σε κάθε χώρα, σε κάθε σύνορο. Επίσης, ε, θα πρέπει το σύστημα να είναι άνετο, να είναι εύκολο να αγοράζει κανείς στήριο, προσιτό και επίσης γρήγορο στην προσφορά που κάνει. Και για τη μεταφορά εμπορευμάτων, επίσης θα πρέπει να πληρούνται οι ανάγκες της αγοράς. Μία από τις σημαντικές προϋποθέσεις είναι η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους για να υλοποιηθεί, για να αναβρεθεί αυτή η ανταγωνιστική ισορροπία και να έχουμε ίσες συνθήκες αγοράς. Γιατί λοιπόν δεν καταφέραμε να υιοθετήσουμε αυτό το σύστημα, γιατί προσκρούσαμε σε διάφορα προσκόμματα που παρεμποδίζουν την εφαρμογή μια επιτυχού τέτοια σιδηροδρομική πολιτική. Για παράδειγμα, ο κατακαιρματισμό του σιδηροδρομικού κλάδου είναι ένα πρόβλημα. Η αργή διάδοση των καινοτόμων τεχνολογιών στην αγορά, αλλά και η πίεση τη αγορά, η χαμηλή πίεση τη αγορά εξαιτία του προστατευτισμού, των επιδοτήσεων των κρατικών και ούτω καθεξής. Και αυτή η χαμηλή πίεση της αγοράς δεν είμαστε σίγουροι θα παραμείνει, γιατί όσο αναπτύσσονται και οι υπόλοιποι εταίροι μας και κυρίως όσο αναπτύσσεται και με ραγδαίους ρυθμούς η αυτοκινητοβιομηχανία, θα δημιουργηθεί περαιτέρω πίεση στην αγορά των σιδηροδρόμων. Ίσως λοιπόν θα έχουμε στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε αυτό, αυτοματοποιημένα βαγόνια που δεν θα χρειάζονται μηχανοδηγό, σειρμούς χωρίς μηχανοδηγό, ή σε ηλεκτρικό σύστημα. Ίσως στο μέλλον λοιπόν θα αναπτυχθούν, θα ανακύψουν πολύ πιο σημαντικές ε, πιέσεις της αγοράς για το σιδηροδρομικό σύστημα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Τώρα, χρηματοδότηση. Και στο παρελθόν αλλά και στο παρόν Έχουμε συγκεντρώσει εδώ κάποια αριθμητικά στοιχεία για να σας παρουσιάσω ορισμένα. 859 ε, δισεκατομμύρια σε επενδύσεις είχαμε στην περίοδο 2000 με 2006 σε υποδομές μεταφορών, σε 25 τότε χώρες μέλη. 112 δισεκατομμύρια από αυτά πήγαν στους σιδηροδρόμους. Και αν δείτε δεξιά, πάνω από το 50% του ποσού αυτού ε, για τους σιδηροδρόμους προήλθαν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση ήταν στο 12%. Ένα μεγάλο τμήμα προερχόταν από μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια ή ιδιωτικά κονδύλια. Αν δούμε τώρα τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης, φτάνουμε σε ένα μακροσκευή κατάλογο ευκαιριών. Ταμείο Συνοχής, το μηχανισμό διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ειδικά Μία και κονδύλια για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Είναι ένα περίπλοκο όμως το σύστημα χρηματοδότησης και απαιτεί πολλές γνώσεις και συμβουλές προκειμένου να συγκροτηθεί μια κατάλληλη χρηματοδότηση για ένα δεδομένο σχέδιο. Οπότε στο μέλλον καλό θα ήταν να, να πλουστεύσουμε κάπως τα πράγματα. Τώρα, στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 διαπιστώνουμε ότι τα κονδύλια που δόθηκαν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για τους σιδηροδρόμους ήταν γύρω στα 82 δισεκατομμύρια ευρώ από το ERDF και το Ταμείο Συνοχής, από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δηλαδή και το Ταμείο Συνοχής και 23,4 δισεκατομμύρια πήγαν στους σιδηροδρόμους, ένα τέταρτο. Και 18 δισεκατομμύρια στις στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και στις υποδομές τους. Στην ε, επόμενη περίοδο προγραμματισμού, για να έχουμε μια συγκριτική κατάσταση, και την περίοδο δηλαδή 2014-2020, είναι 69 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, συν τα κονδύλια από, το, από τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, 24 δισεκατομμύρια. με αντίστοιχο ποσοστό για τους σιδηροδρόμους με αυτό που είχαμε στις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. Ίσως στο τέλος όμως έχουμε κάποια αύξηση των κονδύλιων αυτών ε, από το Ταμείο Συνοχής κυρίως. Για να έχουμε μια μικρή αύξηση σχέση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Σχετικά όμως ανεπέστητη. Οπότε ο πρώτος ε, διαγωνισμός που έκλεισε και αποφασίστηκε στα μέσα του ε, χρόνου είχαμε 14 δισεκατομμύρια για τις μεταφορές και 17, 70% συγγνώμη, από τα κονδύλια αυτά πήγε στο, στους σιδηροδρόμους από το διευκόλυνση συνδέοντος στην Ευρώπη. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό δηλαδή για τους σιδηροδρόμους. Όπως είπα, έχουμε και την πιθανότητα να χρηματοδοτηθούν τέτοια σχέδια από το ΕΦΣΙ, το Σταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δύο δισεκατομμύρια πήγαν από το αρχικά 26 από, το από τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη και δεν ξέρω πόσα θα επιστρέψουν μέσω του ΕΦΣΙ, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, στους σιδηροδρόμους. Αυτό δεν είναι ακόμη σαφές. Είναι σαφές ότι στο παρελθόν είχαμε περισσότερο επενδύσεις σε νέες υποδομές και λιγότερο αποκατάσταση επισκευές. Στο μέλλον θα έχουν περισσότερες τέτοιες επισκευές και αποκατάσταση. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Την ε, ανάλυση κάποιων συγκεκριμένων ε, περιπτώσεων σταθήκαμε σε τέσσερις τέτοιες ε, περιπτώσεις μετά από βιβλιογραφική ανάλυση που κάναμε και εξέταση των εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, κάναμε ανάλυση λοιπόν τέτοιων ε, τεσσάρων τέτοιων περιπτώσεων για σημαντικά σχέδια μεταφορών στην Ευρώπη που έτυχαν και σχετικά προς της χρηματοδότησης. Το πρώτο, τέτοια, το πρώτο τέτοιο σχέδιο είναι η σταθερή ζεύξη του Ερεσούν, που ήταν το σχέδιο προτεραιότητας υπαριθμών 11. Πολύ θετικά τα αποτελέσματά του, γιατί είχε θετικά, θετικό αντίκτυπο και για τις δύο πλευρές. Από τη μια είχαμε το Λούντ και το Μάλμε, από τη σουηδική πλευρά, από τη Δανέζη και την Κοπεχάγη. Και, και μετροπολιτικές περιοχές της Δανίας αλλά και της Σουηδίας ε, εποφελήθηκαν από το σχέδιο αυτό. Για παράδειγμα, οι Δανείοι μπόρεσαν να ε, δουλεύουν στην Κοπεχάγη αλλά να κατοικούν ε, στη Σουηδία. Άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι είδαμε και κάποιες επιπλέον ζεύξεις που αποτέλεσαν από την αρχή τμήμα του σχεδίου. Είναι σημαντικό όταν έχουμε τέτοια μεγαλεπίβολα σχέδια να δούμε και τις επιπλέον ζεύξεις. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε συνδυασμό σιδηροδρομικής και οδικής μεταφοράς. Και μάλιστα ε, διόδια χρησιμοποιήθηκαν ως πόρος για την κατασκευή του σιδηροδρομικού τμήματος. Θα πρέπει να επιτρέπεται τέτοιο, αλλά κάτι τέτοιο προποθέτει και συνδυασμένε υποδομέ οδικές και σιδηροδρομικέ. Άλλη σημαντική περίπτωση υποδομή είναι το τρένο υψηλή ταχύτητα, που συνδέει Παρίσι, Βρυξέλλε, Κολονία, Άμστερνταμ και Λονδίνο. Πολύ θετικό αυτό το σχέδιο προτεραιότητα. είχε πολύ θετικό αντίκτυπο και ωφέλησε κυρίω τα αστικά κέντρα που συνδέθηκαν με το τρένο αυτό υψηλή ταχύτητα και επίσης ε, ωφέλησε για κάποιες ενδιάμεσες πόλεις όπως τη Λίλη στη Γαλλία. Το μειονέκτημα ήταν ότι υπήρξαν κάποιες ε, θεές ζώνες ε, στον Νόρ Παντεκαλέ για παράδειγμα ή στο Κέντ κοντά στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν είχαμε σταθμούς του τρένου υψηλής ταχύτητας οπότε οι περιοχές αυτές δεν ωφελήθηκαν ιδιαίτερα και έμειναν και απομονωμένες. Δεν ε, μπορούσαν να συνδεθούν σε αυτό το δίκτυο. Επίσης είχαμε κάποιες ζεύξεις πρόσβασης ε, και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά όχι αρκετές. Τρίτη περίπτωση, η ζεύξη τρένου υψηλή ταχύτητα ε, στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Για να συνδεθούν η Μαδρίτη και η Βαρκελόνη από την Ιβηρική Χερσόνησο με γαλλικές πόλεις και οι επενδύσεις αυτές ε, ήταν πολύ σημαντικές. Και μάλιστα μερικές φορές ε, εις βάρος των περιφερειακών δικτύων πρόσβασης εξαιτίας των υψηλών επενδύσεων που έγιναν στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας. Ε, η τέταρτη περίπτωση αφορά το σχέδιο προτεραιότητας 22. Τον Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Διάδρομο περνάει από, μέσω Δρέζης από Ορμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Το συμπέρασμά μας ε, για την περίπτωση αυτή είναι ότι ο σχεδιασμός δεν είχε φτάσει σε ένα όριμο στάδιο κάποια τμήματα του διαδρόμου, κάποια κλάδη, ε, το, το τμήμα ε, Πράγας Βουδαπέστης ε, προχωρά καλά, με καλούς ρυθμούς και ο σχεδιασμός φαίνεται προηγμένος και ξεζητημένος, ενώ ο νότιος κλάδος, από τη Βουδαπέστη δηλαδή προς την Ελλάδα, έχει μείνει πίσω. Κάποια τμήματα χρειάζονται καλύτερο σχεδιασμό. Επίσης εξαιτίας των πολιτικών αλλαγών και εξαιτίας της νέας κατάστασης της Σερβίας ε, που είναι χώρα υποψήφια για ένταξη υπάρχει δυνατότητα να ε, εξοικονομήσουμε 300 περίπου χιλιόμετρα ακολουθώντας μια συντομότερη πορεία από τη Σερβία και τη Μακεδονία. Και επίση έχουμε και μια γέφυρα του Δούναβη και άρα συνδυασμό σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και επίση θα βρεθεί χρηματοδότηση από διόδια για προς το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν έχει γίνει. Θα μπορούσε όμως. Και φτάνω τώρα στην τελευταία διαφάνεια Έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας, μιλήσατε 14 λεπτά. Έχουμε στα συμπεράσματα, στα συμπεράσματα για τη συνοχή και την ε, αποτελεσματικότητα της ιδεροδρομικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές, ε, τα διασυνοριακά σχέδια και τα ωφέλη τους, τα ευρύτερα οικονομικά ωφέλη, γενικώ ε, υπάρχουν σημαντικά μακροοικονομικά ωφέλη για τέτοια διασυνοριακά σχέδια. Τα διασυνοριακά σχέδια αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο του σιδηροδρομικού ευρωπαϊκού δικτύου. Αλλά πολλές φορές ε, δεν λαμβάνονται δεν τους υπόψη τις εθνικές πολιτικές. Γι' αυτό και καλό θα ήταν να τα εξετάζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα. Άλλο θέμα αφορά το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας, είναι μια καλή προσέγγιση για τη διασύνδεση των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά χρειαζόμαστε ευρύτερα δίκτυα που θα συνδέονται και με περιφερειακές πόλεις, για να έχουμε πρόσβαση και της περιφέρειας σε αυτό το δίκτυο στο σιδηροδρομικό υψηλή ταχύτητα. Αναφέρθηκα στο σχέδιο προτεραιότητα 22 για τον νοτιοανατολικό σιδηροδρομικό, σιδηροδρομικό διάδρομο στην Ευρώπη, χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων. Και τέλος, τα συμπεράσματα για τα συστήματα και τις μορφές χρηματοδότησης για την πολιτική των σιδηροδρόμων. Υπάρχει περιορισμός σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ιδιωτικά κονδύλια. Μερικές φορές αυτό οφείλεται σε ατέλειες της αγοράς. Για παράδειγμα δεν έχουμε ούτε μερική ούτε ολική εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους, κάτι που πιέζει σε επίπεδο εσόδων, ε, χαμηλή ζήτηση και αβεβαιότητα για τους επενδυτές εξαιτία ε, των, της αλλαγής των προτεραιοτήτων στις πολιτικές. Και επειδή πρόκειται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, η ασφάλεια για τους επενδυτές είναι απαραίτητη. Αν δεν υπάρχει βεβαιότητα για τη μακροβιότητα ενός σχεδίου, τότε δεν είναι ελκυστική μια τέτοια επένδυση, ένα τέτοιο σχέδιο στους επενδυτές. Γι' αυτό και υπάρχει χαμηλό ιδιωτικό ενδιαφέρον. Εξαιτίας λοιπόν αυτής ανεπαρκούς ιδιωτικής χρηματοδότησης με το ισχύον πλαίσιο, υπάρχει ανάγκη να αναζητήσουμε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. Ε, μία λύση είναι το blending, ο συνδυασμός διαφόρων πηγών χρηματοδότησης. Και η ανάμειξη κρατικών κονδυλίων, ε, με κονδύλια ιδιωτικών τραπεζιών ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επένδυσεων ή διαρθρωτικών ταμείων. Αυτός ο συνδυασμός όμως είναι περίπλοκος και χρήζει ειδική τεχνογνωσίας και συμβουλών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από το Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό των ε, της χρηματοδότησης για διάφορα τμήματα, για σύραγγε ή γέφυρες για παράδειγμα. Επίσης υπάρχουν μερικές δυνατότητες χρηματοδότησης για ανάπτυξη νέων συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου για την ανάπτυξη υποδομών. Επίσης, αν δούμε γειτονικέ χώρες, στην Ελβετία για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σιδηροδρομικό Ταμείο και να έχουμε στρατηγικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις για τους σιδηροδρόμους. Υπάρχει κάτι τέτοιο με τους διαδρόμους για τα διευρωπαϊκά δικτύα μεταφορών, αλλά θέλουμε και μια σταθερή βάση για τις χρηματοδοτήσεις που μπορούν να προέρθουν από διαφορετικές πηγές, από τέλη σιδηροδρόμων, από φόρους ε, στα καύσιμα, διόδια και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ, έχουμε τώρα ένα πρόβλημα χρόνου. Ε, είχαμε προβλέψει 15 λεφτά για τις παρεμβάσεις σας και τώρα το έχουμε ξεπεράσει αυτό το όριο. Α, εντάξει. Ε, εντάξει, εάν, ε, εάν δεν θέλετε να αλλάξει το μιλητές το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συντάκτες αυτής της μελέτης, η οποία ήταν μια μελέτη βέβαια για την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και αυτό είχε γίνει με πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και εμείς θελήσαμε να καταλάβουμε από την πλευρά του, της Επιτροπής Ελέγχου του Προεπολεσμού για την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων που δαπανούνται στον τομέα αυτό. Και εδώ θέλαμε να δούμε κατά πόσο επηρεάζει η έλλειψη χρηματοδότησης από τους φορείς τους σιδηροδομικούς ε, στην Ευρώπη για να υπάρξει κάποια βελτίωση. Εμείς πάντως ενδιαφερόμαστε για την ε, χρήση των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη και αυτό το οποίο άκουσα με οδήγησε σε δύο συμπεράσματα. Αν γίνονται διαμεθοριακές ε, επενδύσεις τότε δεν βλέπει κανείς σε εθνικό επίπεδο κάποιο κέρδος. Αλλά αν τα δούμε τα θέματα με ευρύτερο τρόπο, αν τα δούμε κάτω από ένα ευρωπαϊκό πρίσμα, βλέπουμε να υπάρχει κάποια προσθεμένη αξία. Και επίσης πρέπει να δούμε τα θέματα αυτά σε ένα μακρο, πιο μακροχρόνιο ορίζοντα και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μεθοριακές περιοχές πρέπει να έχουν καλύτερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε μια πιο βιώσιμη μορφή επενδύσεων και επομένως ότι ο Σιδηρόδημος πάντα βοηθάει αυτή την αηφόρο ανάπτυξη. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσει κανείς τα ιδιωτικά κεφάλαια. Έχουμε τώρα στο δεύτερο συμπέρασμα της μελέτης όταν μπορέσει κανείς να καταφέρει όχι μόνο να υπάρχουν διαμεθοριακές ε, συνεργασίες αλλά να υπάρχουν και κοινοί φορείς μεταφορών οι οποίοι αναλαμβάνουν την ε, ευθύνη και τον κίνδυνο σε μεγαλύτερες, σε μεγαλύτερες περιοχές. Εγώ βρίσκω πάρα πολύ θετική <clears throat> την ε, διαδικασία στη γέφυρα του Έρεσουν στην Σουηδία και την Δανία όπου οδική γέφυρα χρηματοδοτεί την σιδηροδρομική σύνδεση. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ίσως λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια νέα προσέγγιση στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας τέτοιες ευκαιρίες και να έχουμε μια καλύτερη ε, χρηματοδότηση. Να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό των κονδυλίων και να λέμε πάντα ότι γίνεται μια επένδυση χάρη για ένα οδικό δίκτυο εάν μονάχα παράλληλα γίνεται και μια υποδομή σιδηροδρομική. Πρέπει λοιπόν αυτή η ιδέα να γίνει σαφέστερη σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των ε, μεταφορικών υποδομών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε νέες ευκαιρίες για να <clears throat> βελτιώσουμε την κατάσταση. Σε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά θετικά παραδείγματα, αλλά αν έχουμε μια πιο συστηματική αντιμετώπιση για τα ζητήματα αυτά, μπορούμε να συνδέσουμε με πιο ευφυή τρόπο το ιδιωτικό κεφάλαιο με τα εθνικά κονδύλια και εάν σκεφτούμε τη σημασία των διαμεθοριακών συνδέσεων, τότε νομίζω ότι η μελέτη αυτή πράγματι μας έχει διδάξει κάτι το σημαντικό. Ε, κατακλείδη. Εγώ τώρα δεν είμαι πάρα πολύ καιρό μέσα στην Επιτροπή <clears throat> Μεταφορών, αλλά αυτά που μας παρουσιάσατε με έχουν εντυπωσιάσει όχι μονάχα τα πλεονεκτήματα που παρουσιάσατε, αλλά και τα παραδείγματα αυτά που δείχνουν την επίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο, την δομή της χρηματοδότησης. Αυτό καταδεικνύει πώς λειτουργούν τα πράγματα στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό αυτό είναι μια μελέτη μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και αυτό ήθελα να πω λοιπόν καταλεκτή. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Eh, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, μελέτη που μας παρουσιάσατε. Το βλέπω λίγο με απορία βέβαια γιατί ε, ο τρόπος μέτρησης ε, για διάφορα projects είναι πολύ διαφορετικός. Δηλαδή, με εκπλήσει ότι εσείς εντοπίζετε την πρώτη μελέτη που περιλαμβάνει το Eurostar ως ε, μια επιτυχή ε, υπόθεση. Όμως πάντα έχουμε πρόβλημα με το Eurostar γιατί οικονομικά δεν βγαίνει. Άλλο είναι η συνοχή που εσείς ε, ε, εντάξει το καταφέρνει, το καταφέρνει τη συνοχή, αλλά οικονομικά έχουμε πολλά προβλήματα. Γιατί λοιπόν εσείς ε, και με τι κριτηρία λέτε πως είναι επιτυχής υπόθεση αν λάβουμε υπόψη τα προβλήματα που φέρνουμε μαζί μας συμπεριλαμβανομένου αυτού της χρηματοδότησης. Ιδιαίτερα στο τέταρτο πακέτο ε, το χρηματοδοτικό θα πρέπει να δούμε πώς και κατά πόσο θα περαμείνουν από δοτικά ε, κερδοφόρα ε, τα projects αυτά. Δεύτερον, βλέπω ότι δουλεύετε ε, βασικά με τους επιβάτες. Δεν έχετε κάνει μελέτες με τα εμπορεύματα, φορά εμπορευμάτων. Δεν είδα κατά πόσο δουλέψατε για άλλα τρένα, δηλαδή εκτός αυτά της ψηλή ταχύτητα, και έπειτα για τον διάδρομο του Ατλαντικού και της Μεσογείου με την Νοτιοανατολική, Νοτιοανατολική Ισπανία μάλλον την νότια-ανατολική Ευρώπη, γιατί έχουμε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Τι είναι το δίκτυο, είναι πιο παλιό, είναι κάτι αρνητικό. Και δεύτερον, ο τουρισμός. Άλλες φορές ε, τον υπολογίζετε ως θετικό, άλλες φορές ως αρνητικό. Δηλαδή στις μελέτες που κάνετε τον τουρισμό κάποιες φορές τον βλέπετε θετικά, ενώ άλλες φορές αρνητικά. Άμα θα έχει εδώ πληθυσμός ε, στην Ισπανία θα μειωθεί, αλλά στη Βόρεια Ευρώπη όχι. Λίγο πιο αντιμεγάλη αντικειμενικότητα, τουλάχιστον στον τρόπο με τον οποίο μετράτε, γιατί έχω την εντύπωση ότι σε ορισμένε περιπτώσεις είστε πιο ευνοϊκοί. Υπάρχει δηλαδή ε, αντίφαση στο πώς χρησιμοποιείτε τα ίδια κριτήρια. Εν τω μεταξύ, στο Eurostars εσείς μετρήσατε τα θετικά στοιχεία, ενεργειακή απόδοση ας πούμε, και για το δίκτυο το οποίο ήταν επιτυχές στην Ισπανία που άλλαξε ριζικά ε, η κατάσταση. Εκεί δεν το μετράτε. Αλλά λέτε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και δυσκολίες. Και για την Πορτογαλία θα έπρεπε να πούμε ότι πρόκειται για μια πολιτική απόφαση του, ΕΛΚ, του Λαϊκού Κόμματος της Πορτογαλίας που αποφάσισε να μην το διευρύνει. Και έπειτα το ΕΦΣΙ. Γιατί θεωρείτε ότι είναι τόσο ε, περίπλοκο. Εμείς θέλουμε να είναι συμπληρωματικό της ε, διευκόλυνσης συνδέοντα στην Ευρώπη. Μας ενδιαφέρεται δηλαδή να, να, να μας βοηθήσετε. Ε, δεν μας ενδιαφέρει να μας πείτε ότι θα είναι περίπλοκο, αυτό το ξέραμε. μας πείτε όμως με τις μελέτες που κάνατε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο ώστε να λειτουργήσουν τα πράγματα. Γιατί η διάγνωση που μα ε, παρουσιάσατε ε, μπορεί να είναι αντιφατική γιατί ακριβώ όπω σα είπα διαφορετικά χρησιμοποιείτε τα μέτρα και τα σταθμά και μα είπατε ότι στο νότο δεν θα αναπτυχθούμε άλλο και ότι ο κόσμο θα πάει προ τα βόρεια. Μπορείτε λοιπόν να μου διευκρινίσετε πώς χρησιμοποιείτε τα ίδια κριτήρια για να μετρήσετε αυτές τις ε, περιπτωσιολογικές μελέτες που μας παρουσιάσατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Γκεζίνε. <clears throat> Ο Ντομινίκ και εγώ έχουμε το λόγο και μετά μπορείτε να δώσετε απαντήσεις. Η Γκεζίνε πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της φιλελεύθερης ομάδας θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας παρουσιάσατε. Αναφερθήκατε στην ε, επιτυχία των ε, Ηνωμένων Πολιτειών για τις σύνδεσεις μεγάλων αποστάσεων Έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα βέβαια στις ΗΠΑ, κυρίως μεταφέρουν εμπορεύματα. Τα άτομα πετάνε περισσότερο, δεν χρησιμοποιούν τα τρένα τόσο πολύ όσο στην Ευρώπη. <clears throat> Μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί υπήρξε τέτοια επιτυχία για, το, για τη μεταφορά φορτίων στις ΗΠΑ και ήταν πιο επιτυχές το σύστημα αυτό από ότι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης το θέμα της χρηματοδότησης. Στην αρχή είδαμε με κάπως κριτικό τρόπο αυτό το είδος μικτής χρηματοδότησης, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα για το τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν τα ευρωπαϊκά να χρησιμοποιούνται καλύτερα. Παραγωγή χάρη σύνδεση με την ε, Βουδαπέστη, Αυστρίας Βουδαπέστης είναι ένα παράδειγμα. Τα κράτη-μέλη βέβαια κάνουν την χρηματοδότηση, ξέρουμε τι έχουν κάνει. Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στο θέμα του ιδιωτικού κεφαλαίου που προσπαθούμε <clears throat> να προσελκύσουμε. Έχουμε το Europe Connecting Facility που θέλουμε να βρούμε επενδυτές ιδιώτες για το θέμα αυτό. Τώρα, βλέπω εδώ πέρα να αναφέρεστε σε άλλους πόρους. Αυτοί είναι ιδιωτικοί πόροι και αν είναι ιδιωτικοί ποιο ποσοστό τους Έχουμε το αντιπαράδειγμα βέβαια της ε, Ελβετίας που χρησιμοποιεί κρατική χρηματοδότηση αλλά λειτουργεί ο τομέας αυτός με ιδιωτικά κριτήρια. <clears throat> Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα ο ιδιωτικός τομέας αναλάβει πλήρως την ε, ε, χρηματοδότηση σχεδίων και πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς. Όπως είπατε, θα κάνουν ένα δρόμο να κάνουν και μια συνδρομική σύνδεση. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής της μελέτης. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, με βάση τη μελέτη σας, Μπορείτε να μας εξασφαλίσετε ότι η Κομισιόν διαβεβαιώνει ότι η συγχρηματοδότηση των δύο τελευταίων ετών για τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους αντιστοιχεί στις διατάξεις ε, που είναι σχετικές με την προστεθέμενη αξία που αναφέρεται στον κανονισμό, είτε στο RTT είτε στην διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Μπορείτε να μας δώσετε ένα ε, σωστό παράδειγμα για την συγχρηματοδότηση ε, των διασυνοριακών project όπως ορίζονται στον κανονισμό. Έπειτα, συνάδελφοι, ε, ξέρω θα μου πείτε πως υπερβάλλω και επιμένω σε αυτό το θέμα, η χρηματοδότηση του τούνελ της Βασιλείας ε, της γραμμής Λιών το Ρήνο ανταποκρίνεται στις απαιτήσει διαφάνειας ε, που περιλαμβάνονται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα στη μελέτη σας αναφέρεται το σχέδιο BPK, αλλά αυτό της μεγάλης ταχύτητας το περίφημο, και το αναφέρεται ως επιτυχές παράδειγμα της διασυνοριακής σύνδεσης. Εντάξει, όμως βλέπουμε ότι στις ε, παραδοσιακές συνδέσεις που είναι συχνά διασυνοριακές εκεί εξαφανίζονται. Εξαφανίζονται θα πει τι. Ότι είναι άμεση η συνέπεια όσον αφορά την αύξηση της χρήσης του αυτοκινήτου, άρα αντίκτυπος στο περιβάλλον. Και αυτό σημαίνει πως δεν αντιποκρίνεται καν στην απέτηση που όλοι έχουμε αναφέρει εδώ, τη δέσμευση COP21. Της COP21. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα λοιπόν εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Dominique. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή τη μελέτη που παρουσιάσατε και σήμερα. Έχουμε ήδη ένα πρώτο πρόβλημα και βλέπουμε σαφώς ε, από τις παρεμβάσεις που έγιναν πως αυτή η μελέτη ανατέθηκε από την ΚΟΚΟΜΠΟΥ, την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και όχι από την Επιτροπή ε, Μεταφορών. Α, λοιπόν, βλέπουμε πως ε, υπάρχει μια κάποια δυσαρέσκεια όσον αφορά τα ορίσματα. Αυτή η έκθεση έχει προσανατολισμό τα οικονομικά των project. Πρώτη μου παρατήρηση είναι ε, τι εννοείται results and efficiency. Τι εννοείται. Επί ποιες βάσεις κρίνεται τα αποτελέσματα και την απόδοση των μεταφορών με βάση τη χρηματοδότηση που έχουν λάβει την Ευρωπαϊκή αυτά τα project. Και αυτό είναι ακόμα πιο βάσιμο το ερώτημα γιατί θα πρέπει να σας παραπέψουμε στο πλαίσιο που εν γέννη οι σιδηρόδρομοι οπισθοχωρούν σε σχέση με το παρελθόν ε, και σε σχέση με το μερίδιο της αγοράς. Εάν λοιπόν δούμε ανά ε, μερίδα 100 δις ε, ευρώ, για αυτό το είδος μεταφοράς, τα αποτελέσματα και η δεν ανταποκρίνονται στο ύψος αυτών των χρημάτων. Υπάρχει και άλλη μια ερώτηση που δεν ετέθηκε και θα ήθελα να γνωρίζω αν στην ανάλυση των ευρωπαϊκών θεσμών για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Πάντως ξέρετε γιατί έχουν διαγραφεί οι μεταφορές από τα περιφερειακά μία και από την ανταγωνιστικότητα. Μεγάλη επιβάρυνση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και πώς μπορούν να συνεχίσουν να εξασφαλίζουν τη διασύνδεση <coughs> των γραμμών. Αυτή η απόφαση λήφθη πριν από κάποια χρόνια. Είναι κάτι το οποίο εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε. Έπειτα, οι όροι και η αιρεσιμότητα των ενισχύσεων δεν έχει φανεί, ίσως να μην ήταν και το θέμα όμως της μελέτης αυτής. Έπειτα υπάρχει μεγάλη αριστεία όσον αφορά την ε, ιδιωτική χρηματοδότηση. Το είπατε και εσείς ο ίδιος. Μεγάλη αριστεία εκεί και έπειτα δεν υπάρχει επιστροφή της απόδοσης όσον αφορά τις υποδομές των σιδηροδρομικές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δούμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά και για να δούμε πώς ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να παρέμβει. Πολλές παρεμβάσεις έγιναν, όπου ε, είπαμε ότι ναι, το ΕΦΣΗ με συνθήκες παραπληρηματικότητας θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις δημόσιες επενδύσεις που σιγά σιγά εξανεμίζονται. Εάν όμως θέλουμε πραγματικά να έχουμε την εφαρμογή του ΕΦΣΥ και με την προσθετικότητα θα πρέπει να υπάρχει απόδοση επί των επενδύσεων. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο, υπάρχουν πολιτικά κριτήρια, υπάρχουν κριτήρια διαχείρισης ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας ή απλά και μόνο οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή είναι αποδοτικό, είναι κερδοφόρο, έστω και λίγο το να βάζει κανείς χρήματα στις σιδηροδρομικές υποδομές. Κάτι που είναι πολύ ουσιώδες για τα επόμενα δέκα χρόνια. Τέλος. Και το ανέφεραν και κάποιοι συνάδελφοι. Υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά το τμήμα της ευρωπαϊκής αγοράς και όσον αφορά σε σχέση μάλλον με τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα, την απόδοση, δηλαδή τα εθνικά δίκτυα όπως έχουμε στη Γαλλία και στη Γερμανία που, έχει ε, που έχουμε μονοπόλια ή τις απελευθερωμένες αγοράς υπάρχει διαφορά και ποια είναι αυτή, είναι πολύ σημαντικό. Και έπειτα πέρα από αυτόν τον κατακαιρματισμό των αγορών υπάρχει συμφέρον, υπάρχει ενδιαφέρον στο να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό δίκτυο. Το <coughs> μέγεθος ε, μπορεί να οδηγήσει και σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα ή μήπως οι σιδηρόδρομοι είναι πολύ περιορισμένοι για να ωφεληθούν από συνδέσεις 3.000 χιλιόμετρων ας πούμε ή για να ωφεληθούν από διακρατικές ε, συνδέσεις. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για το μέλλον. τη βλέπουμε το τέταρτο πακέτο για τη διακυβέρνηση θα οδηγήσει σε κατακαιρματισμό των αγορών είναι σοβαρό ή όχι. Θα μας λείπουν τα δημόσια λεφτά. Θα είναι αυτό σοβαρό ή όχι. Είναι δύσκολο να βρούμε και ιδιωτικά χρήματα. Ποια απόδοση μπορούν να έχουν αυτού του είδους επενδύσεις για έναν ιδιώτη. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε μέσα από μια μελέτη για να δούμε ποιο είναι το μέλλον των σιδηροδρόμων. Ευχαριστώ. Να πω κι εγώ κάποια πράγματα. Αναφερθήκατε σε ορισμένα θετικά παραδείγματα όπως αυτό της γεύσης του Ωρεσούντ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν γίνει πραγματικές συζητήσεις όπως για το σύστημα ΦΕΜΕΝ για την συνεργασία των κρατών που θα έπρεπε να συνδεθούν με το σύστημα αυτό. Και δεν υπήρξε η απαραίτητη συνεργασία. Εκεί έχω μια κάποια σκε... κάποιο σκεπτικισμό. Επίσης η ταχεία γραμμή Βερολίνου-Αμβούργου <clears throat> θα ήταν καταστροφή. Ευτυχώς δεν έγινε. Έχει απλώς εξηγιανθεί η υπάρχουσα γραμμή και λειτουργεί μια χαρά. Ή το κανάλι Ειρήνου Δούναβη. Εγώ νομίζω θα ήταν μια μεγάλη βλακεία να γίνει μια τέτοια κατασκευή. Επομένως τα πράγματα είναι πότε είναι καλά τα πράγματα, πότε δεν είναι. Και ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία μπορείτε εσείς να εξασφαλίσετε ότι κάτι θα λειτουργήσει ή όχι. Για την Αδριατική, παραγωγή και τη σύνδεσή τη με τη Βόρεια Ευρώπη, είναι καλύτερα να περάσει κανείς από τούνελ των Άλπαιων ή να περάσει από τι πανονικές πεδιάδες. Και είδαμε <clears throat> ότι στη Γερμανία για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων υπήρξε μια επένδυση 100 ε, δισεκατομμυρίων για την ε, μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων και αυτό δεν είχε αποτελέσματα ουσιαστικά. Ή παραδοσιακά το θέμα του σταθμού της Τουτγάρδης. Για να δώσει κανείς παραδοσιακά στο κομμάτι αυτό του σιδηροδρόμου 10 δισεκατομμύρια για να μειώσει κανείς την, ε, το χρόνο ε, μεταφοράς κατά μερικά λεπτά μονάχα <coughs> ή η σύνδεση με το Βρόσλα, το Βρέσλα ο, ο πρόεδρος. Έχουμε λοιπόν τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη που βλέπουμε ότι δεν προχωρούν τα θέματα αυτά θετικά μέσα στην Ευρώπη. Δεν ενδιαφέρονται φυσικά και όλα τα κράτη-μέλη στον ίδιο βαθμό για να κλείσουν αυτά τα κενά, αλλά η ευρωπαϊκή προστέμενη αξία θα μπορέσει να δημιουργηθεί μόνο αν αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα από κοινού και έχουμε κάποιες, ε, κάποια μελανά σημεία τα οποία θα πρέπει να εξηγιανθούν για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η ευρωπαϊκή προσθέμενη ε, αξία. Δεν πρέπει να σκεφτούμε μονάχα την οικονομική πτυχή, πρέπει να σκεφτούμε και την ανάγκη να προστατεύσουμε την Ευρώπη από την κλιματική αλλαγή, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και γι' αυτό πρέπει να γίνει και η εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια πραγματική αγορά στο μεταφορικό τομέα, είναι ουσιαστικά ένα σύστημα κεντρικού σχεδιασμού σοσιαλιστικής έμπνευσης. Πώς λοιπόν, αυτό είναι όμως το ερώτημά μου, πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε και να εντοπίσουμε τα σχέδια αυτά τα οποία θα έχουν θετικό αντίκτυπο και όχι αρνητικό. Για μένα νομίζω ότι θα ήταν λιγότερο τα μεγάλα ε, σχέδια και περισσότερο τα μικρά σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και έχετε τώρα και οι δύο την ευκαιρία να απαντήσετε. Ευχαριστώ, θα απαντήσω γερμανικά γιατί και εσείς γερμανικά με ρωτήσατε. και ο κύριος ε, Σάντε μπορεί να με συμπληρώσει για τα θέματα αυτά και αυτός φυσικά μπορεί να μιλήσει γερμανικά. Κύριε Κράμερ, ε, τα θέματα της ε, μεταφοράς σε μικρές αποστάσεις δεν έχει τύχει μεγάλης προσοχής. Ορισμένοι τονίζουν την ανάγκη των γραμμών υψηλής ταχύτητας, αλλά η υψηλή ταχύτητα συνδέσει υψηλής ταχύτητας δεν θα πρέπει να παραμελούν και τις ε, τοπικές συνδέσεις, τις συνδέσεις μικρής απόστασης. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε τον διάδρομο ε, Λονδίνου, Παρισίου, Βρυξελών, Φραγκφούρτης. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει αρκετή προσοχή που δόθηκε στις περιφερειακές συνδέσεις και οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα στα Μέρια αυτά δεν έχουν επωφελθεί καθόλου από αυτές τις γρήγορες συνδέσεις. Μόναχα τις μεγάλες πρωτεύουσες ουσιαστικά έχει ωφελήσει το σύστημα αυτό. Αυτό είναι η, το πρώτο, η πρώτη μου απάντηση. Δεύτερον, θα πρέπει να σταματήσουμε να προωθούμε τις ε, συνδέσεις υψηλή Όχι, αλλά πρέπει να δούμε πού είναι εκεί που μπορούμε να συνδέσουμε μεγάλου ε, αστικούς ε, πόλεων και όπου μπορούμε να μεταφέρουμε τον κόσμο από, την, ε, ε, από το αεροπλάνο στο, στο τρένο. Το παράδειγμα του σταθμού της Στουτχάρδης που αναφέρατε. Τα 10 δισεκατομμύρια αυτά τα οποία είχαν δοθεί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για περιφερειακές, για διαμεθοριακές ε, συνδέσει παραδείγματο χάρη μεταξύ Γερμανία και Αυστρία, από το Μόναχο στο Σάλτσμπουργκ και στη Βιέννη. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι υποσυζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά το οποίο μόνο τώρα αντιμετωπίζεται από το Γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών. Θα κόστιζε το 1 δέκατο του σχεδίου για την Στουτγάρδη 2100. Επίσης, υπάρχει πάντα η έννοια της ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας. Αλλά τι είναι η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Είναι σαφές σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Είναι αυτό το οποίο προκύπτει αν ο σχεδιασμός σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να πετύχει πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν σε εθνικό επίπεδο, γιατί τα εθνικά σχέδια φυσικά δεν λαμβάνει υπόψη τις διαμεθοριακές πτυχές. Επομένως πιστεύω ότι μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Δεν έχουμε μονάχα την προσθέμενη αξία σε επίπεδο μεταφορών. Έχουμε την προστασία <clears throat> για το περιβάλλον η οποία μπορεί να προκύψει και την ολοκλήρωση σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Αλλά βέβαια όταν φύγουμε από το καθαρά οικονομικό στοιχείο είναι πολύ πιο δύσκολο να, υπολογίσουμε ποια είναι αυτή η προσθέμενη αξία και εδώ θα πρέπει να είμαστε πιο θαραλέοι να λάβουμε υπόψη μας τις επενδύσεις, το κέρδος σε επίπεδο περιβάλλοντος και σε επίπεδο κοινωνικό. <clears throat> Όπως ελέγχθη, τα αποτελέσματα σε περιφερειακό επίπεδο δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι κάτι που θα γίνει δύο χρόνια μονάχα μετά από την ε, περάτωση μιας επένδυσης. Μπορεί να χρειαστούν 15, 20, 40 χρόνια. Χρειάζεται θάρρος λοιπόν. Δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει όλα και είναι δύσκολο να τα προβλέψει κανείς. Χρειάζεται όμως το θάρρος να δούμε πού υπάρχει δυναμικό και τότε να επενδύσουμε <clears throat> και στο μέλλον. Αν έχω παραδείγματος χάρη ένα σχέδιο τρένου υψηλής ταχύτητας που πηγαίνει στο πουθενά, τότε είναι φανερό ότι αυτό δεν θα έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα σε περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό είναι κλασικό, ότι κάνουμε τις συνδέσεις μεταξύ μονάχα μεγάλων πόλεων και παραμελή τη περιφέρειες, τις περιοχές γύρω από αυτά. Ετέθη το ερώτημα της ε, αποτελεσματικότητας. Τι είναι η αποτελεσματικότητα. Μπορούμε να το ορίσουμε σε οικονομικό επίπεδο, αλλά πέραν του οικονομικού επίπεδου δεν είναι σαφές τι είναι η αποδοτικότητα. Για μένα η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα είναι να μπορεί κανείς να πραγματοποιεί, να υλοποιεί τα σχέδια τα οποία έχει προβλέψει να κάνει. Δηλαδή βλέπουμε τι έχει κάνει, τι προβλεπόταν να κάνει μια επένδυση και ποιο είναι το πραγματικό αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης στην πράξη. <clears throat> και τώρα το ερώτημα αν μπορούν οι σιδηροδρόμοι να φτάσουν αυτούς τους στόχους, πραγματικά τους στόχους που βρίσκονται στις λευκές βίβλες της Κομισιόν, όχι μόνο τους οικονομικούς στόχους αλλά και τους κοινωνικούς και τους περιβαλλοντικούς ε, στόχους, τους στόχους μιας μεγαλύτερης περιφερειακής ολοκλήρωσης. Εγώ νομίζω ότι ο σιδηρόδρομος μπορεί να παίξει ένα μεγαλύτερο ρόλο. Θέλουμε τους σιδηροδρόμους λοιπόν για όλα αυτά ή όχι. Εάν το θέλουμε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερη χρηματοδότηση και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη χρηματοδότηση. <clears throat> και αυτό δεν μπορεί να γίνει μονάχα από ιδιωτικές επενδύσεις. Πρέπει να υπάρξει δημόσια σερμαγιά για να προσελκύσει το ιδιωτικό κεφάλαιο. Μπορούμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, αλλά δεν θα φτάσει. Χρειαζόμαστε και κάποιες εγγυήσει από την πλευρά του δημόσιου τομέα. Πρέπει να υπάρξουν αναλήψεις κινδύνων, εάν θέλουμε να έχουμε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι εύκολο να περιμένει κανείς από τον ιδιωτικό τομέα ε, <clears throat> να συμμετάσχει σε μια διαδικασία που δεν έχει εγγύηση. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να έχουμε μια σύμπραξη, μια κοινοπραξία όπου ο ιδιωτικός τομέας κερδίζει μόνο επειδή υπάρχει η κρατική χρηματοδότηση και εγγύηση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικά. Προσεκτικοί στα θέματα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον το 50% ε, της χρηματοδότησης πρέπει να έρχεται από ιδιωτικό κεφάλαιο. Αλλά υπάρχει και το θέμα του λεγόμενου ηθικού κινδύνου, γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε κάποιους να επενδύουν με την ελπίδα ότι θα καταλήξουν στην τσέπη τους κρατικά κονδύλια. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω δύο πράγματα σύντομα. Το ένα ερώτημα είναι πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη προσαρμογή των σχεδίων στις πραγματικές ανάγκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Παραδείγματος το θέμα της ταχύτητος των ε, τρένων ε, μεταφορικού χαρακτήρα ή η δημιουργία παραλλήλων <clears throat> διάβλων πέραν των ε, βασικών διαδρόμων που έχουμε δημιουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης, όπως είπε και ο προλαλής θα πρέπει να έχουμε και μια διάκριση μεταξύ τη ε, χρηματοοικονομικής απόδοσης, που είναι αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό τους <clears throat> οι επενδυτές, και τη πραγματική οικονομική ε, απόδοσης, άμα λάβουμε υπόψη και όλες τις πηγές εξωτερικού κόστους, που αυτό είναι πιο σημαντικό για τη συνολική οικονομία. Και αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πολύ, και ο πρόεδρο. Κυρία Γιάννη Σάντερ, εκτό μικροφώνου. Είναι πολύ μεροληπτική η παρουσίαση. Μιλάτε ότι με, την, ε, το διάδρομο του Βορρά έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, ενώ με τον Νότο όχι το αντίθετο. Ίσα ίσα. Η προοπτική σας είναι σφαλμένη. Αυτό είπα πριν και δεν το σχολιάσατε. Γιατί το Eurostar το χαρακτηρίζεται επιτυχία με πάνω από 100 υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού, ενώ στο Νότο λέτε ότι δημιουργούνται προβλήματα με το τοπικό πληθυσμό, με τον τουρισμό και το καθεξής. Νομίζω ότι υπήρξε μια παρεξήγηση εδώ. Εμείς δεν επικρινάμε τον τουρισμό. Και τα ίδια μέτρα και κριτήρια χρησιμοποίησαμε για όλες τις περιπτώσεις που αναλύσαμε. δεν καταμετρήσαμε ή δεν αξιολογήσαμε τα σχέδια και τα προγράμματα του Βορρά με διαφορετικό τρόπο αυτά του Νότου. Και μάλιστα το πρώτο σχέδιο που είπατε το ε, που αιρεσούν πούμε, την, ε, το, τη μόνιμη ζεύξη, το αξιολογήσαμε θετικά. Γιατί είναι και οικονομική επιτυχία και επιτυχία διασύνδεσης, αλλά και ο, ε, συμμετοχή των διαφόρων κλάδων, ε, ολοκλήρωση των βιομηχανιών, Δανίας και Σουηδίας, ολοκλήρωση ακόμη και στην πανεπιστημία, σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Και λέμε ότι αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να μεταφερθεί στο Νότο. Είπαμε ότι η Ισπανία επιχείρησε να επιλύσει τα περιφερειακά προβλήματα χρησιμοποιώντας το δίκτυο υψηλής ταχύτητας. Έχει το πυκνότερο δίκτυο στον κόσμο η Ισπανία υψηλής ταχύτητας με τη μεγαλύτερη πυκνότητα ανακάτοικο αλλά έχουν ε, πέντε φορές λιγότερους επιβάτες από ό,τι στη Γαλλία και δέκα φορές λιγότερους επιβάτες από ό,τι στην Ιαπωνία. Άρα δεν μπορούμε να το ε, χαρακτηρίσουμε ως οικονομική επιτυχία με τόσο μικρή ζήτηση. Γι' αυτό ήταν το συμπέρασμα ότι δεν ήταν οικονομική επιτυχία το δίκτυο υψηλή ταχύτητα στην Ισπανία. Ναι, αλλά για τον τουρισμό, για τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Δεν θα σας διακόψω κυρία Αγιάλα Σέντερ. Μπορείτε να τα πείτε σε πηγαδάκι μετά διμερός. Γιατί πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο της της διάταξης. Χωρίς μικρόφωνο κυρία Αγιάλα Σέντερ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συζητητές για τη μελέτη σας. Θα την αναδυθήσουμε με μεγάλη προσοχή. Ganz Ihnen ist es passiert. Λοιπόν, είναι πάντα η δυνατότητα να ε, διευκρινιστούν όλα αυτά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί, να γίνει μια δεύτερη ερώτηση, να διευκρινιστούν τα κτλ. Ερχόμαστε στο πέμπτο σημείο της ε, ημέρας της διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκομένους και με την Κομισιόν για το Uber. Έχουμε τρεις προσκεκλημένους, τον κύριο Μακ Μαγκίν, Μάικλ Νίλσεν και τον Ρομπέρτο Παρίλιο. Οχτώ λεπτά για τον καθένα, ο κύριος Μακ Μαγκίν είναι ο αρμόδιος Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Uber στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ε, ε, χώρες γειτονίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτά, κυρίε και κύριοι, νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ε, έχουμε τετραετή παρουσία ε, στην Ευρώπη, ενώ έχουμε ιδρυθεί εδώ και 5,5 χρόνια. Και μάλιστα δραστηριοποιούμαστε σε 67 χώρες, σε 370 πόλεις, ε, ε, είμαστε σε 23 από τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και μετά τα Χριστούγεννα θα δραστηριοποιηθούμε και σε άλλες τρεις. Τρία εκατομμύρια διαδρομές τον κόσμο, ε, την, την ημέρα έχουμε στον κόσμο, 5 εκατομμύρια το Σαββατοκύριακο και εκατομμύρια οδηγούς στην πλατφόρμα του Uber. Από την ίδρυσή μας αναπτυσσόμαστε και εξελισσόμαστε με γοργούς ρυθμούς και έχουμε δεχτεί πολλά από την εμπειρία μας στην Ευρώπη. Κυρίως δεχτήκαμε από τα παθήματά μας και τα λάθη μας. Πάντως είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της εταιρεία Uber στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να συζητήσουμε πώς νέες τεχνολογίες κινητικότητας με βάση την τεχνολογία οφείλουν και δίνονται να υπο υπαχθούν σε ρύθμιση και εδώ και αλλού. Επίσης, ε, η, η Επιτροπή ζητά ρυθμιστικό πλαίσιο για νέες μορφές ε, κινητικότητας που θα αξιοποιούν τους υπάρχοντες πόρους. Γιατί πριν από πέντε χρόνια τέτοιες υπηρεσίες δεν υπήρχαν, αλλά όλο και περισσότερο χώρες ε, και δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο εξυγχρονίζουν το ρυθμιστικό τους, το κανονιστικό τους πλαίσιο για να επιτρέψουν σωστή ρυθμίση κανονιστική τέτοιων υπηρεσιών που δεν υπήρχαν πριν εφευρεθούν τα έξυπνα κινητά, τα smartphones. Και όπως είπε και η Επιτροπή στο παρελθόν, θεωρούμε ότι ο κατάλληλος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι βρίσκοντας το σωστό κανονιστικό πλαίσιο για να τονώσουμε και να στηρίξουμε την καινοτομία και για την κινητικότητα στις πόλεις. Και γι' αυτό έχουμε συζητήσει με ρυθμιστικές αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί έχουμε μια αγορά με δύο όψεις. Στη μία όψη βρίσκονται οι οδηγοί και στην άλλη οι καταναλωτές. Τα ωφέλη για τον ο, πελάτη είναι εύκολο. Πατάει ένα κουμπί και βρίσκει την σωστή κούρσα. Δεν χρειάζεται να κάνει κράτηση ε, εκ των προτέρων ή να βγει στον δρόμο ελπίζοντας να βρει ταξί. Και όλο και περισσότεροι πολίτες εξαρτώνται από υπηρεσίες σαν αυτές που παρέχει η Uber. Και οι εφαρμογές σαν τη Uber καθιστούν πιο προσιτή και ευκολότερη την πρόσβαση και ασφαλέστερη την κίνηση μέσα στις πόλεις. Ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν έχουν τόσο καλές δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Και παρόλο που πολλές ευρωπαϊκές πόλεις ε, έχουν ε, καλά συστήματα αστικών συγκοινωνιών, πολλές άλλες πόλεις ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα στις αστικές τους συγκοινωνίες. Και αυτή η αυξημένη αποτελεσματικότητα ή αυτή η συμπληρωματικότητα που προσφέρει η Uber, γιατί κατά τη γνώμη μας η Uber δεν προσφέρει Ιού δεν παρεμποδίζει τον υπάρχοντα κλάδο, αλλά συμπληρώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει. Και μάλιστα γίνεται με προσιτό κόστος που ούτε βλάβει τα εισοδήματα των οδηγών. Αλλά διασυνδέει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τους οδηγούς με τους επιβάτες που αναζητούν μια κούρσα. Και έτσι διευκολύνουμε την κινητικότητα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αυτή στα κινητά. Και 70% των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησίας στα smartphones είναι ευρωπαϊκά. Χάρη λοιπόν στην ευρυζωνικότητα, στη δορυφορική πλοήγηση και στα smartphones. Είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη και όστιματα και της επιχείρησης λέω, θα πρέπει να την αξιοποιούμε για οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Και μάλιστα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών και από περιβαλλοντική και από οικονομική και από άποψη μεταφορών. Γιατί έχουμε μια υπηρεσία συνεπιβατισμού. Και ήδη από την δεκαετία του 70 συζητήσατε για αυτή την προσπάθεια κοινή χρησιμοποίηση αυτοκινήτου συνεπιβατισμού, αλλά δεν έχει αποκτήσει τη διάσταση. Στο Σαν Φρανσισκό πάνω από 50% των οδηγών Uber βρίσκονται σε μια νέα υπηρεσία του Uber Pool. Δηλαδή, αντί να έχουμε μόνο ένα επιβάτη με έναν οδηγό, έχουμε δύο, τρει ε, και τέσσερι συνεπιβάτε ε, που ε, χρησιμοποιούν την ίδια κούρσα. Και ενώ ένα οδηγό θα είχε ένα-δύο επιβάτε, τη μέρα τώρα έχει 40 με αυτή την υπηρεσία συνεπιβατισμού. Ε, την περασμένη εβδομάδα ξεκινήσαμε το Uber Pool στο Λονδίνο και έχουμε περίπου 60.000 τέτοιε κούρσες συνεπιβατισμού την εβδομάδα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Οπότε αυτή η διπλή πλατφόρμα ωφελεί και τον οδηγό και τον καταναλωτή. Γιατί με ένα κουμπί έχει κανείς πρόσβαση σε δουλειά ή σε κούρσα. Και μάλιστα οι οδηγοί εταίροι είναι ελεύθεροι για το πότε θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, πόσο θα δουλέψουν ε, και την προσαρμόζουν στη, στον τρόπο ζωής τους και στις ανάγκες τους. Δεν είναι μία δουλειά δηλαδή που ελέγχει τη ζωή τους, αλλά που τους εξυπηρετεί. Και εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο χρησιμοποιούν την εφαρμογή Uber για να οδηγήσουν, είτε ως πλήρη ή ως μερική απασχόληση. Και μάλιστα ως μερική απασχόληση είναι πιο δημοφιλής δραστηριότητα και πιο αποδεκτή στα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. 400.000 οδηγοί χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Uber σήμερα. 50% από αυτούς ε, απασχολούνται λιγότερο από 10 ώρες τη βδομάδα. Δηλαδή το έχουν ως ε, δευτερεύουσα απασχόληση, δεν είναι πλήρης απασχόληση. Στην Ευρώπη που υπάρχει κάποιος κανονιστικός και πολιτικός προβληματισμός έχουμε περισσότερη πλήρη απασχόληση των οδηγών. Και ενώ ε, υποτίθεται ότι θα είχαμε ενιαία αγορά υπηρεσίε βλέπουμε μεγάλο κατακαιρματισμό. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο Έχουμε δραστηριότητες σε 16 πόλεις. 25.000 οδηγούς έχουμε πλήρης απασχόλησης ε, με αδιούχους, επαγγελματίες οδηγούς που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Uber ως βασικό του εισόδημα. Στο Παρίσι έχουμε 12.000 οδηγούς στο καθεστώς ΒΤΣΕ όπως λέμε στη Γαλλία. Μόνο στο Παρίσι και 25% αυτών ήταν άνεργοι προηγουμένως πριν απασχοληθούν στην Uber και 40% από αυτούς ε, θα μπορούσα να έχω χαρακτηριστεί και μακροχρόνια άνεργη πριν βρουν δουλειά στην Uber. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τηρήσω το χρόνο που μου δώσατε. Αυτά προς το παρόν και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες σας. Πάντως ε, ε, θεωρούμε προνόμιο μας αυτή την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων γιατί είχαμε επαφές και με άλλες επιτροπές ε, και η ΤΡΕ και η ΙΜΚΟ ε, το θέμα αυτό στις εξαίσεις για την ενιαία αγορά γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να διαρευνήσουμε νέες οικονομικές δυνατότητες με τεχνολογία και σε καμία περίπτωση να μην παρεμποδίσουμε την πρόοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Μίχαλ Νίλσεν τώρα έχει το λόγο, ο οποίος είναι ο εκπόσωπος της Διεθνούς Ένωσης για τις Οδικές Μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο κύριε Νίλσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμερ, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με προσκάλεσαν <clears throat> για να μιλήσουμε σε ένα, για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ προσφυλές. Η IRU, ερχόμαστε πολλές φορές να μιλήσουμε εδώ για τα θέματα των μεταφορών με φορτηγά, κάτι το οποίο είναι προσφυλές και στον κύριο Κράμερ και εμάς, αλλά και για να <clears throat> εκπροσωπήσουμε τους μεταφορείς με ελευφορία και μεταξύ σε παγκόσμιο επίπεδο. Για μας η οικονομία διαμοιρασμού που χρησιμοποιείται από το Uber και άλλους φορείς είναι τμήμα μιας οικονομίας διαμοιρασμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι μοιράζεται κανείς για να βγάλει λεφτά, μοιράζεται για κοινό όφελος. Αυτό το οποίο κάνει Uber είναι δίνει μεγαλύτερη ε, κερδοφορία σε οργανισμούς και μεγαλύτερη δυνατότητα σε άτομα και επιχειρήσεις. Για μας αυτό είναι ένα θέμα οργάνωσης. Βλέπετε μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο της Μόσχας που λέει προσέξτε <coughs> τους ιδιωτικούς οδηγούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε απάτες και τα λοιπά δεν έχει τα ασφάλεια εξασφαλισμένη. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε κανόνες που θα εξασφαλίσουν ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Όλοι θα πρέπει να σέβονται αυτούς τους κανόνες και θα πρέπει να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός, θεμητός ανταγωνισμός, κανόνες που να ισχύουν για όλους. Και για την Uber. Το να είναι καλή ταξιτζής ή να έχει το σήμα της Uber θα πρέπει να υπόκεινται με στους ίδιους κανόνες αν κάνουν την ίδια δουλειά θα πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες. Αυτή είναι η θέση μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξουν νέοι κανόνες γιατί οι κανόνες υπάρχουν ήδη και πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Δεν θέλετε τους γιατρούς ή τους μηχανικούς ή τους δικηγόρους να, να μην είναι επαγγελματίες. Ούτε θέλουμε να έχουμε οδηγούς οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες και δεν έχουν περάσει μια διαδικασία πιστοποίηση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουν τα εχέγγυα για ασφάλεια, επαγγελματικότητα και τις απαραίτητες κοινωνικές ε, ανάληψη κοινωνικών υποχρεώσεων. Για μας το Uber είναι απλώς ένα κέντρο ουσιαστικά για να μεταφέρει τις πληροφορίες μεταξύ ενός κέντρου και των οδηγών είναι ένα σύστημα το οποίο φέρνει τους οδηγούς των οχημάτων σε επαφή με αυτούς οι οποίοι χρειάζονται να μεταφερθούν, δηλαδή τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν είμαστε οι μόνοι που πιστεύουμε λοιπόν ότι <clears throat> όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μεταφορείς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Αυτή τη στιγμή το Uber λειτουργεί σε 28 χώρες του κόσμου. δεν λειτουργεί σε 28 χώρες, έχει απαγορευτεί σε 28 χώρες. Λέτε στη Γαλλία ότι το Uber λειτουργεί. Αυτό λειτουργήσε μέχρι ότου κάποια από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Uber στη Γαλλία μπήκαν στη φυλακή γιατί λειτουργούσαν με οδηγούς οι οποίοι δεν είχαν άδεια. Και από τότε το Uber δουλεύει με οδηγούς με άδεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να λειτουργούμε χωρίς να σεβόμαστε τους ε, κανόνες. Αν εμείς είχαμε λειτουργήσει στην ε, παγκόσμια οδική οργάνωση όπως το Uber, θα είχαμε βάλει φορτηγά 25 μέτρων σε όλη την Ευρώπη να κυκλοφορούν. Αυτό είναι παραδείγμα των κανόνων, γι' αυτό δεν το κάνουμε. Γι' αυτό εμεί προσπαθούμε να δούμε πώ τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Συνεργαζόμαστε με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας που έχει κάνει μια δήλωση για τα πρότυπα εργοδότησης. Εμείς σε αυτή την κοινή οικονομία, τη διαμεριζόμενη οικονομία, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα ίδια πρότυπα όταν λειτουργεί κανείς παραγωγικά μέσα από το Uber. Υπάρχει ανάγκη να έχουμε κοινέ κατευθυντήρε γραμμέ και ευέλικτε πρακτικέ στην Ευρώπη. Θα πρέπει οι κανόνε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στι ανάγκε των καταναλωτών, γιατί η ταξί είναι τμήμα των δημόσιων μεταφορών. Πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες όλων των πολιτών. Μα τότε πρέπει να εξασφαλίσετε ότι μπορούν να είναι ασφαλής αυτή η υπηρεσία, ότι είναι προσβάσιμη, ότι μπορούν να είναι διαθέσιμοι, ότι μπορούν να παίρνουν χάρη και μετρητά και όχι μόνο αγαπηστοτικές κάρτες. Πρέπει να υπάρχει ισότητα ανταγωνισμού, αλλά πρέπει να υπάρχουν και βέλτιστες πρακτικές. ανέφερε ο Μάρκ, ότι εργάζεται το Uber όπου υπάρχει μια έρημος μεταφορών. Μα για μένα το Uber δουλεύει μόνο στις μεγάλες πόλεις. Εκεί που έχετε ακριβώς τις περισσότερες δυνατότητες μεταφορών. Είναι σαν να μπορεί να νομίζουν κανείς ότι δεν θέλουμε την καινοτομία. Εμείς υποστηρίζουμε την καινοτομία. Εμείς πιστεύουμε στην καινοτομία και στον χώρο των ταξί μέσα στην IRU έχουμε δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο για τα ταξί. Τι σημαίνει αυτό. Θέλουμε να φτιάξουμε καλύτερα ταξί. Όλοι μας είχαμε κακές εμπειρίες με ταξί. Γι' αυτό βλέπουμε τον εαυτό μας ως καταναλωτές και λέμε θέλουμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα. Θεσπίζουμε λοιπόν κριτήρια τα οποία πρέπει να <clears throat> ισχύουν για τις εταιρείε ταξί. Και μετά βλέπουμε τις ε, εφαρμογές για ταξί. Από τότε που ξεκίνησαν τα κινητά τηλέφωνα υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές, αλλά ήταν τοπικού χαρακτήρα. Γιατί αφορούσαν μια πόλη ή μια περιοχή. Αυτό το οποίο λοιπόν γίνεται σε αυτή την περίπτωση είναι απλώς η σύνδεση όλων αυτών των ε, εφαρμογών. Βλέπετε λοιπόν την πράσινη περιοχή όπου είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσει κανείς κάτι τέτοιο και στο υπόλοιπο κομμάτι είναι πιο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διεθνέ δίκτυο με 2,5 δισεκατομμύρια ε, δολάρια, 350.000 ταξί, 1,5 εκατομμύρια ταξίδια κάθε μέρα και αυτό χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια τεχνολογία που υποτίθεται ότι εφήβρε το Uber. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι εμείς δεν προσπαθήσαμε να βρούμε παραθυράκια στην νομοθεσία για να λειτουργήσουμε. Πιστεύουμε ότι όλοι οι πολίτες, όλοι σας, έχουν το δικαίωμα να έχουν ασφαλείς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλα τα μέσα μεταφορών και αυτό περιλαμβάνει και τα ταξί. Αλλά σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα επίπεδο ασφάλειας, ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για τους οδηγούς και αυτό είναι ευθύνη των επιχειρήσεων και τη Uber φυσικά <clears throat> και είμαστε καινοτόμοι στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι υπηρεσίες. Βλέπετε εδώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα, Τέσλα, ταξί Τέσλα. Και αυτά τέθηκαν στη διάθεση ενός καλλιτέχνη ο οποίος έκανε μια εκδήλωση ε, στην περίπτωση αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε καινοτόμοι και να βελτιώνουμε συνέχεια τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ κύριε Νίλσεν. Και τώρα ο κ. Παρίλο από την ε, Οργάνωση Εργαζομένων στις Οδικές Μεταφορές. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, που μας δίνετε την ευκαιρία να εκφράσουμε τη γνώμη μας ε, για αυτό το πρόβλημα στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενδικάτων, Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ε, Οδηγών, την οποία αντιπροσωπεύω εδώ και που είναι παρούσα σε 40 χώρες στην Ευρώπη, είναι μέλος και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων που υπάρχει σε όλες τις χώρες. Θέλω να σας πω το εξής. Είμαστε οπωσδήποτε υπέρ της χρήσης των νέων των τεχνολογιών στην υπηρεσία των πολιτών των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων στο σεβασμό, με σεβασμό στους νόμους που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, εμείς ζητάμε με επιμόνωση η Ευρώπη να χρησιμοποιηθεί ε, για να μπορέσει να υπάρξει ισότιμη στήριξη και μεταχείριση στον τομέα των μεταφορών. Φυσικά όλα αυτά ξεκινούν με την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων. Για παράδειγμα, στον τομέα των οδικών μεταφορών ζητούμε να συγκλίνουν οι πληροφορίες και οι τεχνολογίες που επιτρέπουν ε, να, να ξέρουμε ε, τι ακριβώς σημαίνει, όπως ο ψηφιακός ταχογράφος ε, και ο ευφυής e ταχογράφος για να μπορέσει να υπάρξει ένα ντοσιέ ηλεκτρονικής συμμόρφωσης για όλους τους φορείς. Γαλιλαίο, υγειοεντοπισμός κάθε τρεις ώρες είναι στοιχεία απαραίτητα για να μπορούμε να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό και για να καταπολεμήσουμε κάθε πάτη και κατάχρηση. Κάθε εταιρεία που θέλει να ασκήσει επαγγελματική ε, δραστηριότητα θα πρέπει να σέβεται τους ίδιους κανόνες. Στην Ευρώπη υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός για την πρόσβαση στο ε, ε, επάγγελμα και για την πρόσβαση στη μεταφορά ατόμων επιβατών. Ως μέλη αυτής της Ομοσπονδίας είναι προφανές για μας ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εναρμόνισης και της διοικητικής εναρμόνισης αυτό περνά μέσω της ρύθμισης ε, των ταξί και των ε, νοικιαζόμενων αυτοκινήτων με τα οδηγού στην Ευρώπη. Είτε είναι το Uber, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο φορέα. Είναι απαράδεκτο να ξεκινά την πορεία του στην Ευρώπη μέσω του μη σεβασμού των ισχύων των κανόνων. Πίσω από τις μάσκες με κενά συνθήματα όπως καινοτομία, καλύτερη υπηρεσία στον ε, πελάτη, διαφάνεια, φτύνια, επιπλέον απασχόληση κρύβονται κρύβεται μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Η μεταφορά ανθρώπων από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β δεν έχει τίποτα το κοινοτόμο. Καλύτερη υπηρεσία στον, στον πελάτη για να κάνοντας περισσότερο χρόνο. Διαφάνεια, ας μην το ζητάμε καν, μόλις συζητήθηκε. Φτηνιά, προσιτό, όταν οι τιμές τετραπλασιάζονται από τη μια μέρα στην άλλη, βιώσιμο μια εταιρεία η οποία ζητά από τους συνεργάτες της χιλιάδες ε, να βάλουν ε, ψευδείς ε, παραγγελίες από τους πελάτες. Κάτι ακόμα, μια πρόσφατη μελέτη που έγινε από οικονομολόγους αποδεικνύει το αντίθετο. Η ίδια η έννοια της απάτης δεν έγκυται στο ψέμα το οποίο εκφέρει κανείς, αλλά στην αλήθεια που προτείνει για να καλύψει το ψέμα. Βεβαίως, μπορεί να πει κανείς ότι ο τομέας των ταξί δεν λειτουργεί καλά και ότι το Uber είναι η απάντηση στα προβλήματα. Αλλά αυτό είναι ότι να είναι. Είναι λες και απέναντι σε επικρίσεις που αφορούν το Ευρωκοινοβούλιο θα έπρεπε να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Να σας έλεγε κάποιος ότι πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Ε, όχι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις όταν υπάρχουν προβλήματα σε ένα τομέα. Το Uber απαγορεύτηκε στην Ευρώπη. Αυτό είναι καλό, είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά είναι μόνο το, η κορυφή του παγόβωνου. Το Uber X θα πρέπει επίσης να απαγορεύεται εδώ και καιρό. Ήδη οι δοκιμές για τη μεταφορά εμπορευμάτων και δεμάτων ε, διαφαίνεται στον ορίζοντα. Εκ νέου ε, σε πλήρη άρνηση των ε, ισχύων των κανόνων έχουν εγκατασταθεί στην Ευρώπη αγνοώντας οποιαδήποτε νομοθεσία. Κάθε επιχειρηματίας που σέβεται τον εαυτό του και αποφασίζει να επενδύσει σε μια ε, ε, ε, δραστηριότητα ενημερώνεται. Το Uber κάνει το αντίθετο. Αρχίζει κάνοντας ό,τι του κατεβαίνει περιμένοντας και ε, αποθώντας όλο ένα και περισσότερο τις ε, νομικές ή πολιτικές αποφάσεις που θα του επιβάλλουν να σεβαστεί τις ισχύοντες κανόνες. Ε, οι, Ευρωπαίοι εταίροι των μεταφορών στηρίζουν τις μεταφορές που εγγυώνται τον ενθυμητό ανταγωνισμό, την υπηρεσία στον πελάτη, την ανταγωνιστικότητα της αλυσίδας παντού, το σεβασμό των κοινωνικών και φορολογικών αρχών, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορώ προσωπικά να διαφωνήσω με μια νομοθεσία ή με κάποιον κανονισμό ή κάποια οδηγία και μπορώ να προσπαθήσω να την αλλάξω. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει αυτή η νομοθεσία, ε, καθήκον μου είναι να σεβαστώ τους ισχύοντες κανόνες και αυτό ακριβώς ζητάμε κι εμείς. Να κλείσω δίνοντας ένα ε, συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν ε, σκεφτούμε μια υπηρεσία ταξί και ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό, Όλοι σας μάλιστα, αν έχετε πάρει ταξί στο Ζάβετεν, που σίγουρα θα το έχετε πάρει, πιθανότατα θα έχετε πάρει αυτή την εταιρεία ταξί. Αυτή η επιχείρηση υπάρχει από το 1934. Δίνει ζωή σε 300 οικογένειες και κάθε χρόνο καταβάλει 1,5 εκατομμύριο ε, κοινωνικών εισφορών, 1 εκατομμύριο ε, φόρους ε, και σχεδόν 1 εκατομμύριο ΦΠΑ. Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος ε, πληρώνεται αξιοπρεπώς, καταβάλει τους φόρους του, καταναλώνει, συμβάλλει στην κοινωνική ασφάλιση. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, εφόσον σήμερα είμαστε ασφαλισμένοι έναντι ασθενειών και ατυχημάτων, εάν έχουμε κοινωνική ασφάλιση που λειτουργεί στην Ευρώπη, εάν τα παιδιά μα μπορούν να ακολουθήσουν πανεπιστημιακέ σπουδέ χωρί να χρειάζεται να πληρώνουν τα μαλλιά τη κεφαλή του οι γονεί, εάν έχουμε λοιπόν αυτό το κοινωνικό σύστημα, αυτό είναι χάρη σε αυτό το σύστημα ανακατανομής. Αυτό που το Uber και όλοι οι άλλοι που θέλουν και όλοι οι άλλοι που δεν σέβονται τους ισχύοντε κανόνες θέλουν να εκμηδενήσουν και σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε με κάθε νόμιμο μέσο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτοί ήταν οι τρεις ομιλητές μας σε σχέση με την προβληματική του Uber. Για ορισμένους είναι θαυμάσιο, για ορισμένους άλλους είναι απαγορευτέο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Έχουμε ένα μεγάλο μακρύ κατάλογο ομιλητών. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον. Πρέπει όμως να σας περιορίσω δύο λεπτά οι συντονιστές και ένα λεπτό οι υπόλοιποι. Ο κύριος Φαντερκάπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατρανώνει την επιθυμία της ε, για καινοτομία, για ανατερισμό, για πρόθεση της ψηφιακής αγοράς, της κοινωνίας πληροφορίας. Και όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα φαίνεται ότι δηλιάζουμε μπροστά τους. Ήμπερ, είναι συνεργατική οικονομία, όπως μας είπε κάποιος συνάδελφος. Όχι, δεν είναι συνεργατική οικονομία, αλλά είναι μια προσοδοφόρος ε, μέθοδος και μάλιστα κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Επικερδής δραστηριότητα με ζητούμενο μόνο το οικονομικό όφελος. Επίσης, ε, τι είναι το Uber, παροχή υπηρεσίας ή μεταφορές. Αν είναι θέμα μεταφοράς, είμαστε εμείς ε, αρμόδιοι, αλλά είναι θέμα υπηρεσιών η Επίτροπος Βιενκόφσκα είναι αρμόδια και όχι Επίτροπος ε, για τις μεταφορές. Κύριε Παρίο και Νίλσεν, νομίζω ότι κάποιες ε, μορφές ε, της εφαρμογής Uber θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές. Τι γνώμη έχετε. Κύριε Μαγγέλ, ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του Uber. Γιατί ακούω πολλά και διάφορα. Ακόμη και επαγγελματίε οδηγίε σε ταξί λένε στον ελεύθερο του χρόνου θα ήθελα να δουλέψουν για την Uber. Δεν ξέρω αν στέκουν όλα αυτά. Η Uber εκεί που δραστηριοποιείται, δραστηριοποιείται έχει επιτυχία, αλλά πληρεί τι ε, προδιαγραφέ ποιότητα και τι κοινωνικέ προδιαγραφέ. Δεν θέλουμε ένα αμερικανικό σύστημα χωρί κοινωνικέ προδιαγραφέ. Γιατί είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει υψηλέ προδιαγραφέ και ποιότητα αλλά και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ατυχήματο, Πώ θα διαθετηθεί η κατάσταση. Ο Ισμαήλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, είναι μια συζήτηση αυτή όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν καθαρά τα πραγματικά στοιχεία και όχι απλώς να υπάρχει επιχειρηματολογία η οποία δεν λέει τίποτα το ιδιαίτερο. Θέλω να προκαταλάβω το εξής. Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα και τη λειτουργία της Uber. Εγώ λοιπόν κατανοώ ότι υπάρχουν κατηγορίες κατά τη Uber, αλλά καταρχήν η οικονομία επιμερισμού δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια λανθασμένη ιδέα. Είναι χρήσιμο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ιδέα ακόμα και αν υπάρχει διαφορά με τις ε, παραδοσιακές ε, οργανώσεις ταξιδίδων. Τώρα. Εγώ μπορεί να βρίσκω λοιπόν θετική την υπηρεσία της Uber και ως εκπρόσωπος της σοσιαλιστικής ομάδος θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα στον κύριο Μαγκέν και επίσης στον κύριο Νίσιν και στον κύριο Πάλι. Κύριε Μαγκέν, είναι αλήθεια ότι σας κατηγορούν ότι λειτουργείτε σε μια φαιά περιοχή όπου δεν υπάρχει πραγματική ρύθμιση. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το, αυτή την κατηγορία. Όταν σας λένε ότι έχετε οδηγούς οι οποίοι δεν έχουν άδεια. Δεν πληρώνουν φόρο, δεν έχουν άδεια για ταξί. Τι κάνετε λοιπόν και με τα θέματα ασφάλισης των οχημάτων και των οδηγών. αν γίνει ένα ατύχημα, πληρώνετε εσεί ή πληρώνει ο οδηγό. <clears throat> Όλα αυτά τα ερωτήματα νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε για να έχουμε μια πιο σαφή, μια μεγαλύτερη σαφήνεια και να υπάρξει και μια ευρύτερη <clears throat> αποδοχή από την κοινωνία. Επίσης, ένα δεύτερο ερώτημα. Χρόνο, το χρόνο σας παρακαλώ λέει. Έχετε περάσει ήδη το χρόνο σας. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά τη τα θέματα του περιβάλλοντος. Υπάρχει μια μελέτη από <clears throat> σε ό,τι αφορά το μέλλον της ε, οικονομίας επιμερισμού για τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος. Για τη Νέα Υόρκη, παραδείγματος χάρη, βλέπει κανείς ότι επειδή είναι τόσο φθηνές οι, οι μεταφορές έχουν ανέβει από 14,8 το 2013 σε 17,5 εκατομμύρια μεταφορές το 2014. Τελικά αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος. Και το τελευταίο μου ερώτημα. Υπάρχουν και για τους ε, παραδοσιακούς οδηγούς ε, ε, ταξί γιατί υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί είναι τόσο πολύ εναντίον του Uber. <coughs> Ευχαριστώ. Δύο λεπτά για την για τον επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ. Καταρχήν, περιμένουμε τις δύο μελέτες που ολοκληρώνονται από τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις και φαντάζομαι θα προβαίνουν σε πολύ τεκμηριωμένες αναλύσεις και αξιολογήσεις γιατί οι σημερινές ε, παρουσιάσεις ήταν κάπως υποκειμενικές και νιώθω σαν να είμαι σε δικαστήριο και έκανε σημαντική επίθεση ο κύριος Νίλσεν ήταν πολύ ψηφικά τα επιχείρηματά του γιατί δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε ποτέ ταξί αλλά αυτό που μας είπατε δεν συνάδουν με τη δική μου εμπειρία εγώ προσπαθώ να τα αποφεύγω μετά από εμπειρίες που είχα και, και σίγουρα αυτό που μας είπατε για πολλές χώρες δεν ισχύουν τώρα Κύριε Μαγκάν, πρόκειται για μια νέα επιχείρηση. Σίγουρα υπάρχουν κενά, υπάρχουν παραθυράκια. Θα πρέπει να καλυφθούν τα κενά. Και επίση θέλουμε συνθήκε ανταγωνισμού, δίκε, θεμητέ, ανταγωνιστικότητα, καταβολή φόρων και όλοι να δραστηριοποιούνται επίση όρει. Εσεί κρίνετε την επιχείρησή σας ε, ως ε, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή μεταφοράς. Σε τι κατηγορία εμπίπτεται, στις υπηρεσίες ή στις μεταφορές. Επίσης, προς τους τρεις καλεσμένους θα ήθελα να ρωτήσω. Αυτές οι υπηρεσίες, ας πούμε, αλληλεπικαλύπτονται ή το κοινό είναι διαφορετικό, οι πελάτες είναι διαφορετικοί. Έχετε στατιστικά στοιχεία, γιατί μίλησαμε για φορολογία, για ατυχήματα, Έχετε καθόλου στοιχεία για τα σημεία αυτά και πώς τα βλέπετε. Αυτά βλέπετε. Βλέπω, αρχίζετε και δυσανασχετείτε κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι εξαντλή, έχω εξαντλήσει το χρόνο μου. Σταματώ. Καθόλου δεν νιώθω άσχημα. Κρατήσατε το χρόνο σας και αυτό είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ. Ο κόσμος εξελίσσεται ραγδαία οι πολίτες, οι νέοι πελάτες, οι νέες γενιές. Οι ανάγκες αλλάζουν. Οι νέοι δεν έχουν ε, τις ίδιες ανάγκες με τους πιο ηλικιωμένους. Θέλουν διαφορετικό κόσμο, θέλουν διαφορετικές υπηρεσίες και αν το δικό μας ε, σημείο κίνησης είναι αρνητικό και ε, κατηγορηματικά και μια μονοκοντιλιά απορρίπτουμε οτιδήποτε καινούριο, τότε θα απογοητεύσουμε τους νέους που έχουν υψηλές προσδοκίες από εμά. Θα πρέπει και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουμε μία βάση δραστηριοτήτων που δεν θα περιθωριοποιεί τους νέους ή τους παλιούς. Θα πρέπει όλοι με συνθήκες θεμητού και δίκαιου ανταγωνισμού και σεβόμενοι τους ίδιους κανόνες να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Θα πρέπει φυσικά να γίνονται σεβαστές οι νομοθετικές διατάξεις. Μπορούμε να επιτρέψουμε τις νέες υπηρεσίες ε, ε, οδηγών ε, όπως αυτές προσφέρει η Uber στο κοινό μας. Δεν θα πρέπει να έχουμε αντιπαράθεση μεταξύ παλιών και νέων παρόχων υπηρεσιών γιατί χαμένοι από μια τέτοια αντιπαράθεση και μάχη θα είναι οι καταναλωτές, οι πελάτες σε τελική ανάλυση. Έχουμε λοιπόν νέες υπηρεσίες και έχουμε και πελάτες που θέλουν κάτι καινούργιο αλλά δεν έχουν ακόμη αρχίσει να χρησιμοποιούν τις νέες ε, υπηρεσίες. Ο κόσμος αλλάζει όπως σας είπα. Είμαστε έτοιμοι εμείς για τις νέες αυτές αλλαγές. Θα πρέπει να βρεθούμε στην πρωτοπορία και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει και το θέμα της ε, αμοιβή και της καταβολής φυσικά φόρων για τις δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Κύριε Μαντέλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας και σας ευχαριστώ που είπατε πως η έκθεση της βιώσιμης, η σχέση μάλλον βιώσιμης ε, αστικής κινητικότητας είναι πολύ σημαντική γιατί θέλουμε τη συνδεδεμένη κινητικότητα. Μιλήσαμε για τη νέα γενιά, εντάξει δεν είμαστε και τόσο ηλικιωμένοι, εγώ τουλάχιστον δεν αισθάνομαι τόσο ηλικιωμένη, οπότε να μιλείτε, μιλήσω για την κινητικότητα. Όλοι συμφωνούμε κύριε Νίλσεν, δεν είναι συνεργατική οικονομία το Uber, όλοι συμφωνούν. Αλλά τι είναι τότε, τι είναι το Uber? Είναι μια πλατφόρμα που φέρνει σε επαφή ιδιώτες. Άρα θα πρέπει να πούμε ναι, είναι μια υπηρεσία μεταφορών. Αλλά εκεί έχουμε την εντύπωση πως υπάρχει πρόβλημα, διότι είναι ένα μείγμα των δύο, ναι ή όχι. Εγώ πιστεύω πως είναι ναι, ένα μείγμα των δυο. Και αυτό ίσως μας βοηθά να καταλάβουμε περισσότερο την ε, δραστηριότητά σας κύριε Uber, γιατί στην ουσία μένετε, είστε ένα, μια υπηρεσία μεταφορών, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για εμπορεύματα. Πρέπει να σκεφτούμε αυτή τη δραστηριότητα μέσα στο πλαίσιο της συνδεδεμένης κινητικότητας, γιατί δεν αναγνωρίζεται απλώ λοιπόν ότι πρόκειται για μια νέα επιχείρηση μεταφορική εταιρεία βασικά. Και έπειτα είπε και η συνάδελφοι ένα μαύρο σημείο, δηλαδή το θέμα της φορολόγησης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνισμό και για ηθική μέσα σε πλαίσιο μιας νέας οικονομίας. Εγώ δεν μιλάω για συνεργατική οικονομία, πρέπει να φτιάξουμε μια οικονομία πλατφόρμας. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για την νέα αυτή οικονομία εάν δεν εξετάζουμε από πού έρχονται τα κέρδη και πού πάνε. Μιλάμε συχνά για φορολογικούς παραδείσους, θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και αυτό το θέμα, το θέμα δηλαδή των φόρων. Τρίτον, στοιχεία. Προστασία των στοιχείων, των δεδομένων, όπου σήμερα υπάρχει πρόβλημα, γιατί μιλάμε για νέες τεχνολογίες, ε, αυτά τα δεδομένα που πάνε χέρι-χέρι. Το Uber έχει αποδείξει με, με πιστικό τρόπο ότι μπορούμε, μπορεί κανείς να καταχραστεί τα δεδομένα των ιδιωτών, των προσώπων. Σε αυτό μπορείτε να μου απαντήσετε και έπειτα να έρθω στη δική μου γενιά. Γιατί πιστεύω πως βρισκόμαστε σε μια φάση ε, όπου μπαίνουμε στον 21ο αιώνα, όπου μπορεί να απαγορεύουμε το Uber, αλλά είναι όπως τα ναρκωτικά όπου τη δεκαετία του 20 ε, γίνεται αυτή η προσπάθεια σήμερα ακόμα και αν το σταματήσει κανείς και πει ότι δεν είναι καλό θα γίνει παράλληλη οικονομία. Άρα εμείς ως νομοθέτες τι πρέπει να κάνουμε. Ε, το συμφέρον μας είναι να προβλέψουμε αυτή τη νέα τεχνολογία. Και τελειώνω Πρόεδρε, έχουμε μια ευκαιρία σε αυτήν την Επιτροπή να είτε να νομοθετήσουμε προωθώντας την ψηφιακή ανάπτυξη και ταυτόχρονα <coughs> σεβόμενοι αυτά που είπαμε, τους κοινωνικούς κανόνες κτλ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να είμαστε σε θέση να πούμε ναι, μπορούμε να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε όλοι να ε, συμφωνήσουμε. Ξεπεράσετε κατά ένα λεπτό κύριο Πέτερ Λούντρεν. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σαφής. Νομίζω ότι αυτές είναι μαύρες δραστηριότητες και δεν έχουν καμιά σχέση με την νόμιμη δραστηριότητα του ε, ταξιτζή. Δεν ξέρετε ποιος ε, έστειλε τον οδηγό που σας ε, οδηγεί. Ο οδηγός μπορεί να μην έχει καμία εκπαίδευση, μπορεί να μην έχει το απαραίτητο δίπλωμα, δεν έχετε ιδέα για το ποιος <clears throat> φέρει την ευθένη της ασφάλισης. Τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την παραδοσιακή δραστηριότητα των ταξί στην Ευρώπη. Εσείς κύριε Μακάν, μας λέτε ότι αυτό είναι κάτι το καταπληκτικό. Για την τσέπη σας είναι θαυμάσιο σίγουρα, γιατί εσείς είστε ο κύριος <clears throat> ωφελούμενος από όλα αυτά. Μιλάτε για άνεργους οδηγούς οι οποίοι βρίσκουν δουλειά. Μα ελέγχεται αν αυτοί οι άνθρωποι είναι πράγματι σε θέση και έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αφού είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Το Uber, το επιχειρηματικό του μοντέλο, έχει όλα τα στοιχεία που με κάνουν να είμαι αντίθετος. Αν φέρετε λοιπόν μια τέτοια λειτουργία η οποία βρίσκεται στο πλαίσιο, στο, εκτός του πλαισίου του νόμου, μπορεί αυτή να είναι κερδοφορά. Τι γίνεται όμως με την ασφάλεια, τι γίνεται αν έχει κάποιος ένα ατύχημα, τι γίνεται αν κάποιος τραυματιστεί και μείνει ανάπηρος. Πώς ξέρετε ότι το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιείτε είναι ασφαλές. Ποιος θα ελέγχει αυτά. Πώς ελέγχεται ότι πληρώνονται φόροι. και ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία που πρέπει οι σοβαρές εταιρείες να εφαρμόζουν. Ευχαριστώ. Και τώρα. Οι υπόλοιποι ομιλητέ ξεκινώ με το Κούν. <clears throat> Είναι δύσκολο σε ένα λεπτό, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Η νομοθεσία για τις ε, μεταφορές είναι, κάνει σαφές ότι πρέπει να έχουν και οι οδηγοί της Uber να έχουν τα απαραίτητα ε, πιστοποιητικά. Είναι έτσι ή είναι κάτι το οποίο πηγαίνει οποιοδήποτε ιδιώτης και οδηγεί ένα αυτοκίνητο. Και τι γίνεται με, την τεχνική, με τον τεχνικό έλεγχο. Τα ταξί θα πρέπει κάθε χρόνο να περνάνε ένα έλεγχο, ένα ειδικό έλεγχο. Και πιστεύω ότι αυτό είναι απαραίτητο να ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα τα οποία κάνουν μια τέτοια μεταφορά. η δουλειά του οδηγού χρειάζεται κάποιες γλωσσικές και γεωγραφικές γνώσεις. Επίσης, μπορεί κανείς να διαπραγματεύεται ελεύθερα τις ε, τιμές. Για τη Γερμανία ξέρω ότι υπάρχουν <clears throat> ταρίφες οι οποίες ισχύουν. Τότε μπορεί να κανείς να χρησιμοποιήσει αυτές τις τιμές, αλλά μόνο με τις ίδιες συνθήκες. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Σίγουρα σε αυτό το θέμα θα επανέλθουμε εκτενέστερα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Μία προοπτική που δεν άκουσα ήταν τι γίνεται από άποψη διακυβέρνησης αστικής και τις δυσκολίες που δημιουργείται σε θέματα διαχείρισης του δικού δικτύου, ασφάλειας του δικού δικτύου, αλλά και το θέμα του κανονιστικού πλαισίου. Δεν το σχολιάσατε καθόλου. Επίσης, κάποιες ερωτήσεις. έχουμε πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις που δραστηριοποιείται η Uber και μάλιστα έχουν ασκηθεί πολλές προσφυγές στο Ηνωμένο Βασίλειο για στρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων και χορήγηση μισθών κατώτερων από το κατώτατο όριο. Έχετε λοιπόν ήδη προβλήματα. Ενθαρρύνετε τους οδηγούς με τέτοιες τεχνολογίες να γραφούν ε, και να οργανωθούν σε συνδικάτα, γιατί θέλουμε ένα τέτοιο πλαίσιο. Σε πολλές πόλεις έχουμε κορεσμό από τον υπερβολικό αριθμό ταξί. Γενικώ θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των ε, ταξί, να, τη, χρή, τη χρήση του ταξί για να περιορίσουμε και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Από αυτή την άποψη προς τα που πηγαίνουμε. Ιώζεφ Αμπρί. Ζωζεφ Αρία. Ευχαριστώ κύριε θα ήθελα να πω στον κύριο Παριλιώτ στη χώρα μου, στην Πορτογαλία. Το σύστημα των ταξί είναι αναποτελεσματικό σε ό,τι αφορά την κατάσταση των οχημάτων, την κατάρτιση των οδηγών και επίσης σε ό,τι αφορά το κόμιστρο. Ξέρω ότι υπάρχει ένας κανονισμός στην Πορτογαλία για τα θέματα αυτά των κομίστρων. Η πραγματικότητα είναι ότι οι τουρίστες στη χώρα μου <clears throat> διαμαρτύρονται γιατί δεν εφαρμόζονται αυτά, αυτά τα κόμιστα και οι κανόνες. Για το Uber τώρα. Θα να πω ότι από την πλευρά του καταναλωτή είναι μια υπηρεσία που ισχύει αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία και είναι ευγνώμονες οι <clears throat> καταναλωτές. Αλλά βέβαια πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση και μια σειρά κανονισμών σε σχέση με τη φορολογία, την κατάρτιση την ε, ε, ασφάλεια και τα λοιπά. Αν τα εξασφαλίσουμε αυτά, για μένα το Uber ε, στην Πορτογαλία τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Είναι κάτι το οποίο είναι ακαταμάχητο. Ε, Aiuto. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ήδη είπαν οι συνάδελφοι, σαφώς το Uber είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το μέλλον που μας περιμένει. Όμως θα πρέπει να είναι ένα μέλλον ρυθμισμένο και να προχωρά στην κατεύθυνση που θέλουμε. Δηλαδή να μειωθούν όσο γίνεται τα κόστη για τον πολίτη, αλλά όχι με κάθε τίμημα. Γι' αυτό και έχω κάποια ερωτήματα. Ορισμένα ήδη αναφέρθηκαν, όπως ας πούμε απορίες για τη φορολόγηση, σε ποιον θα καταβάλλονται οι φόροι, σε κάθε κράτο εκεί που λειτουργεί δηλαδή το Uber, δραστηριοποιείται το Uber, μένουν στο κράτο ή πάνω αλλού τελικά απορίες όσον αφορά την ασφάλεια, την εγγύηση, ποιος εγγυάται, πώς εγγυάται το Uber την αξιοπιστία των ε, οδηγών, αλλά και για τα στοιχεία και την ιδιωτική, τον ιδιωτικό χώρο. Πού φυλάσσονται, στην Ευρώπη, στην Αμερική, Ποιοι, ποιος αυτά τα ρυθμίζει αυτά και πώς. Πρόκειται για τεράστιο όγκο στοιχείων. Θέλουμε να ξέρουμε λοιπόν, να γνωρί... Ε, ε, να γνωρί... μπορεί κανείς να γνωρίζει ποιες είναι οι μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών μέσα από αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Σίγουρα θα χρειαστεί να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ τους καλεσμένους και τις πληροφορίες που μας έδωσαν και περιμένω με ανυπομονησία τις δύο εκθέσεις το 2016. Κύριε Μαγκάν. Μιλήσατε για την Uber ως τμήμα της συνεργατικής οικονομίας. Θεωρείστε ε, ότι είστε ψηφιακή πλατφόρμα, πάροχος υπηρεσιών ε, και τι γίνεται με την ιδιωτικότητα των δεδομένων, πώς ελέγχεται ο επαγγελματισμό των οδηγών, τι γίνεται με, τους, με τις αμοιβέ τους, ε, πώς πληρώνονται, πώς αμοιβόνται. Νομίζω ότι χρειάζεται νομοθετική ρυθμίση, γιατί υπάρχει νομοθετικό κενό. Και αν είστε μια ψηφιακή ε, υπηρεσία μεταφορική, θα πρέπει να υπάρχετε σε συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις. Αλλά τι ακριβώς είστε, από πού προέρχεστε και σε τι νομοθεσία θα πρέπει να εμπίπτεται. Νομίζω κάποιο έλεγχο θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Αυτό είναι η βασική μα ανησυχία. Η Uber υπάρχει, είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε πια να την αναχαιτήσουμε και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Και πολλοί καταναλωτές χρησιμοποιούν την εφαρμογή αυτή με τα κινητά τους. Δεν ξέρω σε τι βαθμό, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον θα πρέπει να ικανοποιήσουμε τους καταναλωτές, συμπληρώνουμε τα νομοθετικά κενά. Κύριε Σινίλσεν, Ευχαριστώ. Η υπηρεσία Uber μέσω της εφαρμογής είναι προσιτή παντού στην Ευρώπη και στη Σουηδία. Αλλά στη Σουηδία όλοι πληρώνουν φόρους και για την δραστηριότητα αυτή. Μερικοί όμως που χρησιμοποιούν την εφαρμογή σας κατέληξαν στα δικαστήρια. Έχουμε 20 τέτοιες ε, αγωγές κατά της Uber και μάλιστα η, η νομολογία χαρακτήρισε τις ε, υπηρεσίες της Uber ως ε, εμπορικές δραστηριότητες και μάλιστα αντίθεται στην Σουηδική νομοθεσία. Η Uber λοιπόν είναι παράνομη στη Σουηδία. Δημιουργήθηκε όμως ένα παραθυράκι και χωρίς να έχετε καμία υποχρέωση, χωρίς ε, να πληρώνετε κανένα φόρο, παρέχετε υπηρεσίες. Και όταν η εφορία μας ανακαλύπτει τους οδηγούς, τους υποχρεώνει να πληρώνουν φόρους. Αλλά εσείς ως εταιρεία θα πρέπει να λάβετε τις ευθύνες σας. Γιατί έχετε διαπράξει απάτη σε μεγάλο βαθμό. Κριστίνα Αρνούτο. <coughs> Είπε κάποιος ότι τα έσοδα του Uber μπορούν να αντιμετωπίσουν την ανεργία. Εδώ είναι λοιπόν το δίλημα. Κάποιοι θέλουν την απόλυτη φιλελευθεροποίηση του, των υπηρεσιών και της μεταφοράς με τρόπο που πολλές φορές μπορεί να είναι αθέμητα. Μια άδεια οδηγού ταξί μπορεί να κοστίσει 200.000 ευρώ. Και από την άλλη πλευρά θεωρούμε ότι ένα κράτος θα πρέπει <clears throat> να δώσει τη δυνατότητα να έρθουν τα νέα επαγγέλματα στην, στην επιφάνεια και να έχουν την κατάλληλη οργάνωση. Αυτό το οποίο γίνεται με το Uber ε, έχουμε το πρόβλημα ότι πολλές φορές πολλοί οδηγοί οι οποίοι είναι άνεργοι κάνουν μια μικροδουλειά, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό ε, πρόσθετο εισόδημα. παραμένει μια δραστηριότητα η οποία είναι επισφαλής και μερικού χρόνου. <clears throat> Πιστεύουμε ότι τα κυρίαρχα κράτη θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια ρύθμιση για το θέμα αυτό και όχι να γίνει με μια ευρωπαϊκή ρύθμιση η οποία θα οδηγήσει σε κινδύνους και νομικούς αλλά και φορολογικούς γιατί μπορούμε να έχουμε εταιρείε οι οποίες δεν πληρώνουν το φόρο στις χώρες όπου λειτουργούν. η Κριστίνα Βονταλόν. Ευχαριστώ τουλάχιστον στη Γαλλία μία ε, εναρμόνιση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Κομισιόν έχει καταλάβει πως υπάρχει μια σύγκληση απόψεων από πλευρά των συναδέλφων σήμερα στο ότι η καινοτομία θα πρέπει να ωφελήσει όλους τους φορείς μεταφορών επιβατών. Αλλά οι κοινωνικοί, οι φορολογικοί οι κανόνες και οι κανόνες ασφάλειας και ευθύνης θα πρέπει επίσης να εναρμονιστούν. Δεν γίνεται δηλαδή να έχουμε δύο διαφορετικά μέτρα και στάθμα. Είναι επίγον λοιπόν να υπάρξει αυτή η εναρμόνιση ε, για, τα, ε, ε, όλα τα θέματα, για την υγεία, την σύνταξη, την αδιαμητρότητα, θέματα ασφάλισης, ένα σωρό ζητήματα που εάν δεν υπάρξει εναρμόνιση του συνόλου των μεταφορέων επιβατών δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και αυτή η καινοτομία δεν θα μπορέσει να ωφελήσει όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Στη συζήτηση αυτή νιώθω σαν να βρισκόμαστε στη δεκαετία του 50. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν ε, είχαμε ε, εισαγωγή του rock and roll από τις Αμένες Πολιτείες και στην Ουγγαρία ε, οι επιτροπέ των οδών του Σοβιέτ συνεδρίαζαν για το κατά πόσο θα το επιτρέψουν ή όχι. Νομίζω ότι από συζητήσει με ταξιδίδες στην Ουγγαρία μαθαίνει κανεί πολλά. Και οι συνάδελφοι με κοροϊδεύουν όταν παραπονιέμαι για τις κακές υπηρεσίες που προσφέρουν οι ταξιδιδε και στην πατρίδα μου και στις Βρυξέλλε. Και πολλοί συνάδελφοι με συμβουλεύουν να αφήσω το ταξί και να χρησιμοποιώ οδηγού στη Σούμπερ. 25 ε, εκατομμύρια πολίτες ε, είχαμε στη δεκαετία του 50. Τώρα έχουμε πάνω από 100 εκατομμύρια τουρίστες που διακινούνται συνεχώς. Οπότε και χάρη στις ψηφιακές ε, υπηρεσίες πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάπτυξη και, την, και της τεχνολογίας αλλά και του τουρισμού. Θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Μίχαλ Γκάλερ. <clears throat> Πρέπει να πω καταρχήν ότι εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμα ποτέ το Uber. Έρχομαι από τη Φραγκφούρτη, πηγαίνω με το ταξί στο αεροδρόμιο. Και δεν ξέρω πόσα μένουν σε ένα ταξιτζί ο οποίος τηρεί όλες τις προδιαγραφές. Μου λένε οι ο οδηγός ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν στην μαύρη για ένα ποσό κατά αποκοπή και ουσιαστικά ανταγωνίζονται τα επίσημα ταξί. Γιατί, Γιατί για πολλούς ανθρώπους το ταξί είναι πολύ ακριβό <clears throat> και γι' αυτό υπάρχει αγορά για το Uber. Και ιδίως στις πόλεις που δεν υπάρχει καλή δημόσια, καλές δημόσιες μεταφορές. σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης μπορεί κανείς να κινείται καλά με τις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά είναι άλλες περιοχές στο, Ιου, στο πούμε, μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ουσιαστικά δημόσια συγκοινωνία και ο κόσμος παίρνει το Uber γιατί οι ταξιτζίδες είναι διεφθαρμένοι και ακόμα λιγότερο αξιόπιστοι. <coughs> Στη δεκαετία του 90 είχα πάει στην ε, Πράγα και μου είπανε μην πάρεις ταξί γιατί είναι όλοι ύποπτοι και διεφθαρμένοι. Μπορώ να καταλάβω λοιπόν ότι κάποιοι χρησιμοποιούν το Uber γιατί είναι φτηνότερο λοιπόν και πιο βολικό και πιο ασφαλές. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια λύση για όλα αυτά τα θέματα. Είναι μια, θα πρέπει να είναι μια λύση που θα εξασφαλίσει ότι όλες αυτές, όλα αυτά τα δικαιολογημένα αιτήματα των ταξιτζήρων θα μπορέσουν να γίνουν ε, να γίνονται δεκτά. Η Ισαμπέλ. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να κάνω, να καταλαβαίνω μάλλον ότι είναι ένα, μια ζήτηση και βρίσκει μια προσφορά. Όμως όταν ε, κάτι είναι ρυθμισμένο είναι ε, καλύτερα. βέβαια, μπροστά σε αυτό το δίλημα, το πώς να βρούμε εδώ μια λύση, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο νομοθέτης ε, θα πρέπει να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον. Ασφάλεια και πληρωμή των ε, συνεισφορών, αλλά και βέβαια ισότιμη μεταχείριση όλων. Άρα λοιπόν ποιο είναι το κριτήριο κατά τη γνώμη μου. Όταν υπάρχει οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα πρόκειται για μια επιχείρηση. Η επιχείρηση έχει κόστος, ε, έχει ασφαλιστικές συνεισφορές, φορολογικές εισφορές, γραφειοκρατικές υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Θα ήταν λοιπόν ε, θέμα πολιτικής να βρούμε κίνητρα για τις ζώνες που δεν εξυπηρετούνται τόσο πολύ από τις δημόσιες υπηρεσίες ή για τις ε, περιοχές όπου υπάρχουν ανάγκες που σχετίζονται με μια μερική υπηρεσία να διευκολύνουμε, αλλά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι ο γνώμονας ή ισότητα μεταχείριση, ίση μεταχείριση. Θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς ποια πιστεύετε θα είναι η ισοτητα ή θα ηθελα να ρωτησω ρύθμιση στο sharing economy, στο πλαίσιο του sharing economy. Έβαλα Το εαυτό μου στο τέλος του κατάλογου. Αν είναι παρακαλώ και εσείς. Περίμενα κι εγώ τη σειρά μου. Ε, βρήκε ευκαιρία η Uber να αναπτυχθεί, γιατί και οι ταξιδίδες υπάγονται στην περίφημη επικουρικότητα, που είναι γενικώ καλή, αλλά μερικές φορές είναι κακή όταν ήταν ήδη καλή η τοπική ρυθμίση. Βρήκε λοιπόν κενό και χώθηκε η Uber. Πάντως, όντως, μπορεί να είναι εύκολο να πατήσει ένα κουμπί και να βρει ταξί, αλλά το κάνουμε αυτό ήδη στη Μαδρίτη, στην πατρίδα μου, δεν είναι μόνο η Uber που έχει προσφέρει τέτοιε τόσο προσιτέ υπηρεσίε και οι ταξιδιώτε είναι οργανωμένοι και μπορεί εύκολα κανεί πατώντα ένα κουμπί να βρει ταξί. Ερωτώ λοιπόν την Uber. Για πόσα μένουν από κάθε κούρσα στην Uber, πόσα πληρώνει στην εφορία και πότε, και πού μάλλον, συγγνώμη. Επίσης, ε, τι ευθύνη έχει η Uber απέναντι στους επαγγελματίες ή στους οδηγούς, γιατί δεν είναι όλοι επαγγελματίες. Δεν είναι σίγουρο αν έχουν άδεια οδήγηση ή άδεια ε, οδηγού. Υπάρχουν πολλές νομικές πτυχές που είναι πολύ σημαντικές ε, στην παροχή ε, μεταφορικών υπηρεσιών. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας, πόσο είναι ασφαλισμένος ο οδηγός, τι γίνεται σε περίπτωση ατυχήματος ή σε περίπτωση που αρρωστήσει ο οδηγός, τι ευθύνη θα αναλαμβάνει απέναντι στο πελάτη η Uber. Επίσης, τι γίνεται με την ιδιωτικότητα των στοιχείων. Τι κάνει η Uber με τα δεδομένα ε, αυτών των ε, μεταφορών. Ευχαριστώ. Για μένα το ταξί αφορά τις ε, κοντινές διαδρομές και έχω μιλήσει πολλές φορές με τους ταξιτζίδες μου έχουν πει ότι, ε, ότι είναι πολύ φθηνότερε οι τιμέ τη Uber. Αν κάνει κανεί λοιπόν την απαραίτητη κατάρτιση, άμα εξασφαλίσει τον ελάχιστο μισθό για του οδηγού Uber και έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλές ε, επιχειρήσεις οι οποίες είναι απατηλές. Συνέχεια, ε, αλλάζουν τα, τα δεδομένα των χιλιόμετρων πολλές φορές οι εταιρείε για να κερδίσουν πιο πολλά λεφτά. Όταν είμαι στο αεροδρόμιο και θέλω να πάω δύο χιλιόμετρα, μου λέει ο ταξιτής δεν πάω γιατί αυτό η κούσα μου δίνει μονάχα 5 ευρώ. Περιμένω μια ώρα εδώ πέρα στο αεροδρόμιο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Γιατί δεν μπορώ να έχω ένα ταξί σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ε, ανταγωνισμό, αλλά πρέπει να είναι θεμητό ανταγωνισμός. Θα δώσω λοιπόν το λόγο σε αντίστροφη σειρά πρώτα στον κύριο Παρίγιο. Μάλιστα. Δεν θα ακρηγορήσω. γιατί κάνετε μια πολύ καλή ανακεφαλαίωση της κατάστασης. Οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για όλους. Ο θεμητός ανταγωνισμός, ο ισότιμος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σε αυτή την αρχή στηρίζεται, αλλά δυστυχώς αυτέ τις αρχές δεν τις σέβεται η Uber. Και αν δεν φροντίσουμε, καταπάτηση τέτοιων αρχών θα γίνει και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Ή λοιπόν θα κάνουμε μια επιλογή. Λέμε ναι στην καινοτομία, στον εταιρισμό, στις νέες τεχνολογίες, αλλά προσοχή. Όπως είπε και παρακαθήμενος, θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ της συνεργατικής οικονομίας και του business. Γιατί είναι σημαντική η ορολογία που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε όποια και αν είναι η επιχείρηση, η Uber, η Α ή Β επιχείρηση, όποια επιχείρηση και αν είναι, να σέβεται τους ισχύοντες κανόνες. Και αν δεν υπάρχουν κανόνες, αν υπάρχουν κενά, να θεσπίσουμε κανόνες. Για ε, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι η στρατηγή της επιχείρηση Uber δεν είναι να αρχίσει να ενημερώνεται για τους ισχύοντες κανόνες, είναι να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες μέχρι ότου μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια ή η πολιτική ή δικαιοσύνη θα επιβάλλει στην Uber κανόνες ε, απορρίπτοντας τον ένα ή άλλο τρόπο μεταφοράς. Έχουμε μια χιονοστιφάδα νεοτερισμών που αυτή τη στιγμή όμως βρίσκονται στην παρανομία ακόμη θα πρέπει να απαντήσει μια πλούστατη ερώτηση η Uber. Είναι πρόθυμη να τηρήσει τους κανόνες που πληρούν και οι υπόλοιπε επιχειρήσεις. Ναι ή όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον ζήτημα και περιμένω την απάντηση του, της Uber γιατί μέχρι στιγμής λέει όχι στους χιόντες κανόνες και αν η απάντηση είναι όντως όχι θα πρέπει να λάβουμε δραστικά μέτρα. Ο Μιχαήλ από την IRU. Θα προσπαθήσω εγώ να απαντήσω σε όσο το δυνατόν περισσότερα <coughs> ερωτήματα. Ο κύριος Άτρουκ είπε ότι είναι καλή ιδέα η βασική σύλληψη για το Uber. Και εγώ συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να γίνει μέσα στους κανόνες, με σεβασμό των κανόνων και δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και γι' αυτό πρέπει να αντιδράσουμε. Ναι, φάνηκε σαν να ήμασταν σε ένα δικαστήριο. Ναι, γιατί στα μέσα ενημέρωση και μεταξύ των πολιτικών φαίνεται ότι τα λεφτά μιλάνε τα εκατομμύρια, τα εκατο, εκατοντάδες εκατομμυρίων των, της Uber έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες εξαρτήσεις των μέσων ενημέρωσης για να στρέψουν το κοινό υπέρ του Uber. Και δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αλλαγές. Μα υπάρχει νομοθεσία. Λειτουργήστε μέσα στην νομοθεσία ή αλλάξετε την νομοθεσία. Νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε τα πράγματα καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Και ρωτήσατε αν είναι διαφορετικοί οι πελάτες. Όχι, οι πελάτες είναι. <clears throat> τα ταξί κάνουν πράγματα που δεν τα κάνει το Uber. Μεταφέρουν ανθρώπους που είναι ανάπηροι. Μεταφέρουν ανθρώπους σε αραιοκατοικημένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν ελεοφορία ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά μπορούν να πάρουν τους ανθρώπους εκεί που θέλουν να πάνε, μπορούν να πάνε τους ασθενείς στα νοσοκομεία έξω από τις μεγάλες πόλεις. Υπήρξε ένα ερώτημα για την ε, Uber. Τι είναι Uber, είναι μια υπηρεσία που στέλνει ταξί στον πελάτη. Επομένω είναι μια μεταφορική υπηρεσία, επομένω πρέπει να υφίσταται την ίδια ρύθμιση. Κύριε Λούντγκεν, είχα καιρό να ακούσω σου ειδικά. Για μένα είναι σαφές ότι η Uber δεν έχει καμία αστική ευθύνη. Λέει στα ψηλά των, των ε, προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα ε, του θα δείτε ότι αποσύουν οποιαδήποτε ευθύνη, οποιαδήποτε αστική ευθύνη για αυτό που κάνουν. Για την Πορτογαλία. Και εγώ είπα ότι όλοι μας έχουμε εμπειρία από κακές υπηρεσίες ταξιτήρων. <clears throat> και εγώ πολλές φορές βρίσκομαι στο αεροδρόμιο και δεν με παίρνει κανένα ταξί και αναρωτιέμαι. Γιατί. Αυτό δεν είναι εντάξει. Θέλουμε να αυξήσουμε όλη την ε, βελτίωση, να βελτιώσουμε την ποιότητα. Αυτό δεν είναι θέμα νέων νόμων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι μεγαλύτερη την ε, ε, ποιότητα. Και στην Πορτογαλία υπάρχει μια υπηρεσία με app που σου δίνει και την τιμή οπότε δεν μπορεί να σε κλέψει ο ταξιτζής. Και αυτό μπορεί να γίνει με τα νόμιμα ταξί. Για τα συνδικάτα μπορείτε να μου απαντήσετε, λέει η κυρία Άντερσον. Ναι, θα το έλεγα τώρα αυτό. Για μας, ο, η επιχείρηση του ταξί θα πρέπει να λειτουργεί μέσα στο νόμο αν είναι υποχρεωμένοι να έχουν μια συμφωνία με τα εργατικά συνδικάτα, ναι, πρέπει να το κάνουν. Και θα πρέπει να σέβονται τις συλλογικέ συμβάσεις όπου υπάρχουν. Αυτό είναι προφανές. Αν είναι κανείς ε, σύνομος, θα πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό υπάρχουν οι κοινωνικοί εταίροι και διαπραγματεύονται για να καταφέρουν τις καλύτερες αυτές ε, συνθήκε. Αυτά. Και Σα uh, Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής για τις ε, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Δεν είμαι βέβαιος πόση ώρα μου δίνετε. Πέντε λεφτά, γιατί μετά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Δεν θα απαντήσω ατομικά σε κάθε αν και θα είδατε ότι έγραφα με τα μανία. Νομίζω όμως ότι ε, σημείωσα τα πιο και κύρια σημεία από αυτά που αναφέρατε. Και αν δεν το έκανα, αν δεν απάντησα, παρακαλώ να μου ξαναρωτήσετε. Είμαι ευτυχής που καταρχήν που το Ευρωκοινοβούλιο ε, μα έχει καλέσει. Ήμασταν προσκεκλημένοι διαφόρων πολιτικών ομάδων παλιότερα. Τώρα είναι η πρώτη φορά που η ίδια Επιτροπή μας ζήτησε να έρθουμε και να πούμε τη γνώμη μα. Ε, παρά να εξαρτάται από διάφορες ε, ε, εκθέσεις. Και φυσικά θα ξανάρθουμε οποτεδήποτε ε, χρειαστεί. Είμαι ευτυχής που η συζήτηση δεν στρέφεται γύρω από το αν θα γίνει το Uber, αλλά πώς θα γίνει το Uber. Και εδώ δεν είναι μόνο το Uber, βέβαια. Είναι για κάθε νέα οφειή τεχνολογική εταιρεία που θέλει να κάνει μια επιχείρηση είναι το πιο, το πιο οικείο. Και το πιο είναι το Airbnb. Υπάρχουν και διάφορες άλλες νεοφυείς, όπως BlaBlaCar και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες. Σε ιδιαίτερα στην μεταφορά επιβατών ε, στις ασταστικά κέντρα, οι κανόνες που ισχύουν, οι νομοθεσίες που ισχύουν δεν ε, αντιστοιχούν, γιατί αυτά έγιναν στην βιομηχανική, για τη βιομηχανική κατάσταση. Τώρα είμαστε στην τεχνολογική ψηφιακή εποχή και θα έπρεπε οι σχετικές νομοθεσίες να προσαρμοστούν. Ξέρω ότι δεν είμαστε σε δικαστήριο, αλλά ε, θέλω να σας παρακαλέσω όταν καλείτε κόσμο να τους ζητάτε αυστηρά να έχουν και πρακτικές ε, ε, αποδείξεις, γιατί κάποια από αυτά που υπόθηκαν δεν είναι ε, σωστά, δεν είναι, δεν είναι αληθή. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν, είπε η κυρία Κούν, Είστε κάποια πλατφόρμα, είστε μια νεοφυής, είστε συνεργατική οικονομία, sharing economy ή collaborative economy όπως το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα αν είμαστε μεταφορική εταιρεία ή ψηφιακή πλατφόρμα, όχι, εμείς λέμε ότι είμαστε ψηφιακή πλατφόρμα. Οι υποδομές υπάρχουν, υπάρχουν οι τηλεπικοινωνίες και οι, το, με, δορυφόρων πρόκειται για μια αυξανόμενη ομάδα ε, επιχειρηματιών του λογισμικού και βασιζόμαστε σε υπάρχουσες ψηφιακές δομές. Δεν είμαστε λοιπόν μεταφορική εταιρεία. Μέχρι το τέλος του 2016 ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα σας πει μια και έξω αν αυτό είναι μεταφορές, είναι ψηφιακή υπηρεσία ή είναι κάποιο υβρίδιο. Πάντως αυτό θα πρέπει να καθυστερήσει την εκπόνηση της νομοθεσίας για την χορήγηση άδεια. Όπως είπα υπάρχουν δύο ειδών Uber για τους ιδιώτες ε, οδηγούς 25.000 ε, Λονδρέζοι αυτή τη στιγμή ε, δουλεύουν με αυτή την κατάσταση. Βγάζουν το ψωμί τους έτσι. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί που δουλεύουν στα μαύρα τελείως. Το Ηνωμένο Βασίλειο, κοιτάξτε, υπάρχουν και 90.000 ιδιωτικά αυτοκίνητα όμως σε μεταφορικές εταιρείες. Εγώ μπορώ μόνο να μιλήσω για το Uber. Πάντως είναι ένα καθεστώς που είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Ε, το άλλο άκρο είναι η Ισπανία που απαγόρεψε το Uber. Ε, σημαίνει πως 50.000 κόσμος που το χρησιμοποιούσε καθημερινά δεν μπορεί πια να το χρησιμοποιήσει. Τώρα, όσον αφορά τη χορήγηση ιδεών, έχετε το καθεστώς VTC στη Γαλλία. Όπως είπαν, ε, θα σας πούν η κυρία Ντέλ και η κυρία Ριβό, όμως είναι δίκαιο να ζητάμε από κάποιον ε, να μελετήσει για 250 ώρες, ενώ όταν πρόκειται για ελαφρά αεροσκάφη μόλις 25 είναι υποχρεωτικές ώρες ε, ε, πτήσης. Είχαμε το Uber Pop που εξακολουθεί να υπάρχει σε κάποια κάτι μέλη. Δεν απαγορεύτηκε στις 28 χώρες αν η ασφάλιση δεν καλύπτει ατύχημα, αυτό που κάνουμε είναι ότι καλύπτουμε το 1% που μπορεί να συμβεί. Ε, το Uber έχει μια γενική πολιτική ασφάλισης που ε, ε, υπερασφαλίζει το αυτοκίνητο του οδηγού υπό το γαλλικό ή βελγικό ότι είναι υποχρεωτικό να έχει κανείς εμπορική ασφάλιση. Τώρα για τη φορολόγηση. Η φορολόγηση ομίλων, Το 80% των όσων δαπανά στο Uber ε, πάει στον ίδιο τον οδηγό. Είναι νομική υποχρέωση του κάθε οδηγού να καταβάλει τη φορολόγηση, είναι συμβατική του υποχρέωση και όπως είχε αναγνωρίσει και η κυβέρνηση της Γαλλίας, η οδηγοί του Uber είναι στην ουσία independent, self-employed, ανεξάρτητοι επαγγελματίε. Εάν λοιπόν κανεί αμφισβητήσει το δικαίωμα να είναι αυτεπάγγελτο, να είναι μάλλον ανεξάρτητο επαγγελματία, τι πρέπει να κάνεις, να πληρώσεις τις κοινωνικές σου εισφορές, αλλά δεν μπορείς να αμφισβητείς το δικαίωμα της Uber να χρησιμοποιεί την ε, ψηφιακή τεχνολογία σε, αυτό το, σε αυτή την πλατφόρμα. Όσον αφορά την εμπορική φορολόγηση, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κέρδη. Ελπίζουμε πως κάποια στιγμή θα έχουμε κέρδη. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσον αφορά την εταιρική ε, φορολόγηση ε, και αν αλλάξουν οι σχετικοί κανόνες φυσικά και θα συμμορφωθούμε και στο μέλλον. Άρα λοιπόν είναι άδικες αυτέ οι επικρίσει. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα και τις δημόσιες μεταφορές. Το Uber θεωρεί ότι λειτουργεί συμπληρωματικά. Το 50% των διαδρομών είναι μιας ε, κατεύθυνση. Χρησιμοποιούν δηλαδή άλλο ε, είδος δημόσιας μεταφοράς ή μεταφοράς εν γέννη για να επιστρέψουν. Το Uber πάει στα 200 μέτρα από τη στάση του μετρό, ας πούμε, στο Παρίσι. Αν το δούμε ως μια υπηρεσία κινητικότητας, και νομίζω ότι όσοι, προήλθαν, όσοι μίλησαν από τη Φιλανδία το γνωρίζουν αυτό, πρέπει να δίνεις στον καταναλωτή μια επιλογή. <clears throat> επιλογή είναι δημόσιες μεταφορές, είναι το ταξί, που έχει λαμπρό μέλλον μπροστά τη και υπάρχει το Uber και υπάρχουν ένα σωρό άλλε υπηρεσίε. Ε, ε, ε, δηλαδή, το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να δώσει τα κίνητρα στον κόσμο να αφήσει το αυτοκίνητό του σπίτι του. Δεν ανταγωνίζεται για φόρους, αλλά όχι ανταγωνίζεται την ανάγκη να έχει κανείς ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο, ένα για ταχύ. Ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε θα δώσω και πάλι το λόγο στην Κομισιόν. Ο κύριος Λίζιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σας και λίγο πριν τα Χριστούγεννα να ξεκινήσω με κάτι θετικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η συνεργατική οικονομία μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα αυτό ισχύει και για τις μεταφορές. Με την ανάπτυξη νέων μορφών κινητικότητας. Μπορούν να δημιουργηθούν λοιπόν πολλές ευκαιρίες ε, συνεργατικής οικονομίας προς όφελος των καταναλωτών που θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες, ποιοτικές υπηρεσίες, με θεκτικό αντίκτυπο και στις τιμές. Η συνεργατική οικονομία, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών, μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες και σε, στο επίπεδο της καινοτομία και της απασχόλησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλη αυτή οι πάροχοι των ε, υπηρεσιών θα πρέπει να έχουμε μια ευκαιρία να διεισδύσουν στις εθνικές αγορές. Επίσης όρις όμως με τους ε, ήδη υπάρχοντες παρόχους υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να άρουν τα εμπόδια στην ε, παροχή δραστηριοτήτων ε, και να περιορίσουν τα εμπόδια. Οι νέε αυτέ ω υπηρεσίε δημιούργησαν και κάποιε προκλήσει, ακόμη και ένταση σε μερικέ χώρε μέλη. Έχουμε μάλιστα λάβει πολύ διαφορετικέ απαντήσει από τι εθνικέ αρχέ. Οι παραδοσιακοί κλάδοι υπηρεσιών θεωρούν ότι η Uber δεν πληρεί του ίδιου κανόνε ό,τι αφορά την πρόσβαση στι υπηρεσίε. Πολλά ερωτήματα έμειναν απάντητα σε θέματα ασφάλισης, ε, φορολογίας για παράδειγμα και απασχόλησης σε ό,τι αφορά την Uber. Οπότε, τι κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά. Θα υιοθετούσα μια πολύ ε, συνετή και επιφυλακτική προσέγγιση, γιατί είμαστε ακόμη σε φάση συγκέντρωση πληροφοριών. Δεν έχουμε ε, απόλυτα αποκρισταλωμένη γνώμη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Πάντως, από φιλοσοφικής απόψεως δεν θα πρέπει να ξεχνούμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Καταρχήν θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για νέες υπηρεσίες, ώστε τέτοιες νέες υπηρεσίες να βρίσκουν τη θέση τους στην αγορά. Και επίσης είναι σημαντικό να εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνθήκες ισότιμου και θεμητού ανταγωνισμού. Και με αυτά τα δύο σημεία θα ολοκληρώσω έχουμε ξεκινήσει την εκφώνηση μιας μελέτης για να δημιουργήσουμε καλύτερη άποψη για την αγορά και τις κανονιστικές ρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Δεν είναι μια μελέτη που θα καταλήξει σε νομοθετική πρόταση, δεν έχει το χαρακτήρα μελέτης επιπτώσεων. Στόχος της μελέτης είναι να διαμορφώσουμε μια καλή εικόνα ε, της κατάστασης στην αγορά και της ε, νομοθετικής ρυθμίσης στα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Μερικοί μάλιστα μίλησαν για εξασφάλιση συνθηκών ισότιμων ανταγωνισμού και εναρμόνιση των κανόνων πρόσβασης στο επάγγελμα. Δεύτερη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά την στρατηγική μας για την ενιαία αγορά που εγκαινιάσαμε στις 28 Οκτωβρίου. Και στην στρατηγική αυτή στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής έχουμε αναγγείλει ότι θα δώσουμε κατευθυντήρες γραμμές για την εφαρμογή υπάρχουσας νομοθεσίας προκειμένου να καλύψει και τις νέες αυτές υπηρεσίες της συνεργατικής οικονομίας. Δηλαδή, ε, εφαρμογή ισχύουσας νομοθεσίας σημαίνει οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για τις υπηρεσίες ή αρχές ε, της συνθήκης, ε, ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ελευθερία εγκατάστασης ή θέματα συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία ή τη νομοθεσία για τις ασφαλίσεις. Και μάλιστα, αν διαπιστωθούν από τις μελέτες αυτές νομοθετικά κενά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποκλείται να υποβάλει και νομοθετικές προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με διαφορετικές και ενδιαφέρουσες απόψεις. Φυσικά συνεχίζεται η συζήτηση, αλλά Θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι εμείς υποστηρίζουμε την καινοτομία, αλλά υποστηρίζουμε και τον θεμητό ανταγωνισμό. Θα πρέπει να είναι οι ίδιες οι συνθήκες για όλους και γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που συνεχίζεται. Η Κομισιόν είπε ότι δεν έχει ακόμα αποκρισταλωμένη θέση, αλλά ε, η Ευρώπη θα πρέπει να βρει μια λύση για τα θέματα αυτά γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών, μπορεί να υπάρχουν διαμεθοριακές μεταφορές. Δεν μπορεί η Ευρώπη να λειτουργήσει λοιπόν με διαφορετικά καθεστώτα, πρέπει να έχουμε με ένα κοινό καθεστώς. Συζήτηση συνεχίζεται. Ευχαριστώ την, ε, τους προσκεκλημένους μας και όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο από την Επιτροπή μας. Πάμε τώρα στο σημείο 6 για την ε, απαλλαγή για τις ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Κομισιόν.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 Έχουμε καθυστερήσει λιγάκι, θέλω να συνεχίσουμε. Έχουμε τον ε, συντάκτη γνωμοδότηση τη Επιτροπής μας, τον Μασιμιλιάνο Σαλίνη, για, τον, για την απαλλαγή για τον Γενικό προπολογισμό. Είχε το λόγο. Λυπάμαι. Φοβάμαι ότι θα είναι κάπως λιγότερο ενδιαφέρουσα η παρέμβασή μου από τη συζήτηση που προηγήθηκε. Θα προσπαθήσω να σταθώ μονάχα στα βασικά στοιχεία και να είμαι σύντομο σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του 2014. Πρόκειται για ένα σύνολο για μια σε τρία ε, δις και για τις πληρωμές έχουμε μια υποδιέρεση υποδιέρεση ανάλογα με το κεφάλαιο των μεταφορών των ίδιων που συμπεριλαμβάνουν και τον μηχανισμό του ασφάλειας ε, των επιβατών ε, και των οργανισμών που περιλαμβάνουν περίπου το 80% των, υποχρε... Ε, πληρωμών, υποχρεώσεων πληρωμών. Έχουμε επίσης την καινοτομία, το ΣΕΖΑΡ, έχουμε ακόμα 8% και 6,5% για τις ε, πληρωμές και κλείνουμε με τις διοικητικές δαπάνες ε, όσον αφορά τις 7 και το 7 και το 4. Ε, Τώρα για να περάσουμε γρήγορα στις γραμματοτήσεις που δόθηκαν για αυτή την απαλλαγή. Το ποσοστό εκτέλεσης των υποχρεώσεων αλλά και των πληρωμών είναι εξαιρετικό. Έχουμε 98,2% για τις υποχρεώσεις και 95,2% για τις ε, πληρωμές. Όμως ε, δεν μπορέσαμε ε, παρά να εκφράσουμε μία απογοήτευση για το υψηλό ποσοστό σφάλματος στον τομέα της ανταγωνιστικότητας ανάπτυξης και επασχόλησης, όπου το ποσοστό 5,6% σφάλματος οφείλεται κυρίως στην παρουσία αποζημιώσεων για κόστη τα οποία θεωρήθηκαν μη παραδεκτά. Γι' αυτό και τονίσαμε ότι θα πρέπει να γίνουν εξάντε έλεγχοι όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται αυτό το ποσοστό σφάλματο. Υπάρχει και άλλο ένα σημείο που είναι το 4 στο σχέδιο γραμμοδότησης, όπου ακόμα και αν δεν είμαστε ακόμα στο πια στο 2014, ο Γιούνκερ είναι εδώ και έχει έτσι καταλάβει ένα μεγάλο τμήμα της συζητησή μας στο θέμα αυτό όσον αφορά την σύσταση του προϋπολογισμού στο 2016 που μάλιστα εντός του οποίου η δική μας γνωμοδότηση χεμένα ε, εισηγητή. Χρειάστηκε λοιπόν να καλύψουμε το μέγα θέμα ανάμε, ε, ε, των σχέσεων ανάμεσα στο ΦΕΙΣ και στο ΕΣΕΦ και κυρίως την ανάγκη να διατηρηθεί ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων που θα απευθύνεται στις επενδύσεις. Το ΣΕΦ είναι ένα ε, μέσο, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε λειτουργεί πολύ καλά και γι' αυτό δεν μας άρεσε που διαπιστώσαμε ότι σε κάθε προπολογισμό ένα σωρό προγράμματα μεγάλη, πολύ ποιοτικά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΦΕΙΣ λόγω έλλειψης πόρων, γι' αυτό και εδώ θερήσαμε να βάλουμε μία αναφορά στο σημείο 17 της διαθεσμικής ε, διοργανικής συμφωνίας όπου ζητάμε ευελιξία για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους πόρους που απευθύνονται σε αυτήν ακριβώς του είδους τις επενδύσεις και συγκεκριμένα το ε, ΣΕΦ. Μπορούμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε με ακρίβεια κάθε φάση προόδου των διαφόρων προγραμμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των project τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τον προπολογισμό της Ένωσης που ε, ε, στόχο έχει τις μεταφορές. Υπάρχουν όμως τρία τρεις βάσεις δεδομένων. Έχουμε το σύστημα διαφάνειας, οικονομικής διαφάνειας, έχουμε το ΙΝΕΑ και το Κόρτις για το ορίζοντα 2020. Θέλουμε να δούμε μια απλοποίηση ε, ώστε στο τέλος να έχουμε μία μόνο βάση δεδομένων όπου να απλοποιηθούν οι επαληθεύσεις ε, και οι έλεγχοι ε, τη υλοποίησης αυτών των projects που είναι θέμα κλείδι έπειτα. Έχουμε και αυτό το project Shift to Rail. Ε, ε, Επίση, τονίζουμε το θέμα του τουρισμού που μιλάμε για 11 δις 6,5 για τις υποχρεώσεις και τα υπόλοιπα για τις πληρωμές και πάλι θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν μεγαλύτερο έλεγχο και περισσότερο διακρίδια ε, για τις δαπάνες για τον τουρισμό. Και εν πάση περιπτώσει καταλήγουμε στο ότι θέλουμε να δοθεί απαλλαγή για αυτόν τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή Ευχαριστώ, ευχαριστώ και για την ε, συντομία σας η κυρία Αγιάλα Ευχαριστώ. Εδώ και αρκετό καιρό που ασχολούμαστε με το ελεκτικό συνέδριο. Πρώτη φορά το ελεκτικό συνέδριο δεν υπέβαλε γνώμη επιφυλάξεις για τους οργανισμούς. Οπότε και οι τρεις οργανισμοί συν τον ΣΕΣΕΡ είχαν ανεπιφύλακτη αξιολόγηση. Πολύ καλή είδηση αυτή. Επίσης, οι Ευρωπαίοι, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απαλλαγή και για το shift to rail που είχε ένα πρόβλημα κατά την εκκίνησή του. Αλλά μια και μόνο τον Ιούλιο του 2014 υπογραφτήκε η συμφωνία, δεν ε, μπορέσαμε να δώσουμε την απαλλαγή σε μια αυτόνομη ε, επιχείρηση. Το αφήνουμε για το χρόνο ώστε να τεθεί σε ισχύ το shift to rail. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό για την, την Ασφάλεια σε Αέριες Μεταφορές, εδώ υπάρχει μια σύγκρουση αρκετά σημαντική και καλό θα ήταν να την διαθετήσουμε γιατί τώρα με το συντηροδρομικό πακέτο έχουμε την ευκαιρία για ανανέωση της νομικής βάσης και αφορά την συμφωνία για την έδρα με τη χώρα προέλευσης, ε, προκειμένου τη Γερμανία. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Είχαμε μεταφορά σε άλλο κτίριο και κάποια προβλήματα γιατί ο Οργανισμός Ασφάλειας Αεροπορίας δεν έχει καταφέρει ακόμη να συμφωνήσει με τη Γερμανία για το θέμα του κτίριου. Ενώ η γερμανική κυβέρνηση κατέληξε σε απόφαση το 2011 για την αντίστοιχο οργανισμό για τις ε, επαγγελματικέ συντάξεις και τις ασφάλειες είναι πιο σημαντικέ οι συντάξει από την ασφάλεια στην αεροπορία. Εντάξει, δεν θα επεκταθώ, ούτε θα κάνω α, χαριτολογήματα για το θέμα αυτό. Πάντως, ακόμη έχουμε μια προσωρινή συμφωνία προβληματική, γιατί το ελεκτικό συνέδριο το επισημαίνει. Δεν έχει υπογραφεί ακόμη συμφωνία με την γερμανική κυβέρνηση. Οπότε, όταν στο αεροπορικό πακέτο θα ασχοληθούμε και με τον Οργανισμό ασφάλεια Αεροπορίας, θα πρέπει να σταθούμε στο σημείο αυτό πρέπει η γερμανική κυβέρνηση να δεήσει επιτέλους ε, να υπογράψει τη συμφωνία αυτή με, για την έδρα με, την, με τον Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας. Και μάλιστα έχουμε αναθέσει πολλές προκλήσεις και νέα καθήκοντα στον Οργανισμό Ασφάλειας. Ε, εγκρίναμε και αύξηση του προσωπικού Οπότε νομίζω ότι αξίζει αυτός ο οργανισμός ασφάλειας αεροπορίας ε, μια οριστική συμφωνία με τη γερμανική κυβέρνηση. Δεύτερον, έμψε ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα. Σε μερικές περιπτώσεις ε, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης ε, μετά τα ατυχήματα που είχαμε στη Μεσόγειο και χρειαστήκαμε τη βοήθειά της. Κάποια προβλήματα απομένουν στον οργανισμό αυτό, αλλά ίσω σημασία και χάρη της διαφάνειας που μας είναι προσφυλής, ζητούμε να δημοσιευθούν τα βιογραφικά των υψηλά εισταμένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Για να αποκατασταθεί η διαφάνεια και να διευθετηθούν ε, προβλήματα ή να αποσοβηθούν αμφιβολίες ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων την ενδεχομένη. Σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ των πιστώσεων, η, Ευρωπαϊ... Επιτροπή Ελέγχου προπολογισμού ε, παραπονιέται συνεχώς για το πλεόνασμα που έχουν κάποιοι οργανισμοί. Σε μερικές περιπτώσεις τα πλεονάσματα αυτά οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί ή όχι την πρόσβασή του στον μελλοντικό προπολογισμό και έτσι δημιουργούνται κάποιε καθυστερήσει. Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα υπήρξε πρόβλημα και με το πρόγραμμα για τα σκάφη που κόλλησε κάπου και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί υπήρξε χρεοκοπία της ε, εταιρεία. Αλλά δεν θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει πρόβλημα με τις κυρώσεις γιατί το ελεκτικό συνέδριο πάλι θα επισημάνει προβλήματα. Γιατί υπάρχει μια θεά ζώνη σε ό,τι αφορά ε, τα προβλήματα που θα πρέπει να αναλάβει, ε, να επιλύσει η επιχείρηση που χρεοκόπησε. Τώρα, για τον ΕΡΑ, τον Ευρωπαϊκό Σιδηροδομικό Οργανισμό. Θα αυξηθούν οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του και εξακολουθεί να ταλανίζεται από κάποια προβλήματα εξαιτία κάποιων διαγωνισμών, κάποιων δημοπρασιών. Θεμότητα στο θέμα αυτό θα ήθελα να μα εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται με την πρόσληψη του προσωπικού. Γιατί δεν μπορεί να προσελκύσει ακόμη ιδιαίτερα ειδικευμένο προσωπικό. Και επίση και το θέμα τη σύγκρουση συμφερόντων. Να αποσοβηθούν όλες οι αφιβολίες να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει σύγκρουση φερόντων. και να ξέρουμε από πού προέρχεται το προσωπικό, οι επαγγελματίε. Σίγουρα χρειαζόμαστε ειδικευμένο προσωπικό, να ξέρουμε από ποιες εταιρείες προήλθαν αυτοί οι άνθρωποι και χάρη διαφάνειας θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πάντα για αυτούς. Και σε ό,τι αφορά την κοινή επιχείρηση ΣΕΣΑΡ, αυτή τη φορά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και στο δεύτερο διαγωνισμό είχαμε βελτίωση των οικονομικών συνθήκων. Και ξεπεράσαμε την αρβαιότητα που υπήρξε κάποια στιγμή για την πορεία που θα ακολουθήσει το σχέδιο, η επιχείρηση αυτή και θα μπορούσε να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς τα κατάφερε και το ξεπέρασε, γιατί φαίνεται ότι πραγματικά είχαμε μια καλή λύση. Και όπως είπε και το ελεκτικό συνέδριο, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα όντως έχουν πάρει τη σωστή πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βιμ Φαντακάμπ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μας μένουν 19 λεπτά, νομίζω. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω. Από την πλευρά του ΕΛΚ. Δεν μας ενδιαφέρει <clears throat> το θέμα των ε, αριθμητικών στοιχείων, αλλά το θέμα των ουσιαστικών συμβολών των φορέων αυτών. Η Επιτροπή Ελεύθερου Προϋπολογισμού Προπολογισμού πρέπει να κοιτάξει τα αριθμού, αλλά εμεί θέλουμε να δούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των ε, αποκεντρωμένων φορών. Έρχομαι στους φορείς αυτούς. Σεζάρ, πρώτα απ' όλα. Ο... Η μάνατζερ για την ε, ε <clears throat> ανάπτυξη των συστημάτων και το FES, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για, την, ε, για τις στρατηγικές επενδύσεις. Τι γίνεται σε σχέση με αυτά τα θέματα στο ΣΕΖΑΡ. Τρίτον, πώς επηρεάζει το ΣΕΖΑ τις διάφορες περιοχές. Έρχομαι στην ΕΑΣΑ μετά. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που γίνονται στην ΕΑΣΑ. Μας είπανε ότι είχε μεγαλύτερη ανάγκη για προσωπικό. Έχουν αυξηθεί σημαντικά τα καθήκοντα της ΕΑΣΑ. Το ερώτημά μου είναι αν είναι δυνατόν με το τωρινό προσωπικό να φέρουν σε πέρα σε αυτά τα καθήκοντα. Η ΕΡΑ, η Υπηρεσία για τους Ιδιοδρόμους. <coughs> πόσα χιλιόμετρα από το νέο δίκτυο έχουν ε, δημιουργηθεί. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να δούμε την απόδοση αυτών των υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ, λέγει ο πρόεδρος. Ο Ντομίνικ Κρικέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχά το έφερε ο εισηγητή του Γενικού Προπολογισμού σου και εισηγητή για του Οργανισμού. Να υπογραμμίσω το γεγονός ότι 18 μήνες μετά από την ε, Shift to Rail εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Είναι σκάνδαλο αυτό. Αυτή η παρατήρηση έγινε από τον συνάδελφο Σαλίνη και βέβαια δεν υπάρχει έκθεση βέβαια από την πλευρά των οργανισμών γιατί δεν υπάρχει. Γιατί δεν λειτουργεί. Είναι περίπλοκο, είναι η διαδικασία. Ε, είναι ένα <coughs> πρόβλημα που πρέπει οπωσδήποτε να εγκαλέσουμε την Κομισιόν. Και είναι ζήτημα γιατί όχι μόνο δεν λειτουργεί, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα λειτουργήσει ούτε καν στο επόμενο εξάμεινο. Δεύτερη γενική παρατήρηση, κάτι που υπογραμμίστηκε για τους οργανισμούς, ότι δηλαδή ε, ε, κατά πόσο είναι συμβατό το να αυξάνουμε διαρκώς τα καθήκοντά τους ενώ κάθε χρόνο μειώνουμε τις θέσεις. Είναι καθόδες το ζήτημα και όσον αφορά τις, ε, την ΕΑΖΑ δεν είναι κατανοητό το 90% των πόρων να είναι εκτός του ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού του ίδιου. Δηλαδή να μειώνουμε τις δαπάνες για τις οποίες δεν δίνουμε καν τους πόρους. Ή, εν πάση περιπτώσει, δίνουμε πολύ μερικού ε, τα, τα, κονδύλια. Κάτι ακόμα. Ο τουρισμός είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτής εδώ της Επιτροπής και ο προϋπολογισμός του. Και υπήρξε και έκθεση. Ε, καταλαβαίνετε ποια είναι η σημασία του τουρισμού στην οικονομία μας. 7 με 8% τουλάχιστον του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, 11 εκατομμύρια ευρώ μόνο για προπαρασκευαστικά project χρόνια ε, ε, ζητάμε από την Κομισιόν πρόταση δημοσιονομική που να στηρίζει τον τουρισμό και παραμένουμε σε γελία επίπεδα. Δεν δίνουμε κανένα μέσο για κάτι το οποίο ε, ανέρχεται στο 7-8% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και είναι και μέσα στις συνθήκες. Πρέπει αυτό να το τονίσουμε σε επίπεδο του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Τελείωσα. ο κύριο Φαρία και ζητώ συγγνώμη που δεν τον είδα προηγουμένω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να συγχαρώ την συγγήτρια για τι τέσσερι αυτέ γνωμοδοτήσει. την Αγιάλα Δεν έχω το χρόνο να διεξέλθω μεμονωμένα κάθε μία από αυτές τις γνωμοδοτήσεις. Θα λάβω το λόγο συνολικά για όλες αυτές και θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της ΕΜΣΑ, που είναι αυτή που γνωρίζω καλύτερα. Την... Έχω προσωπική γνώμη, έχω πάει εκεί και φυσικά εδράζεται στην δικιά μου πόλη, στη Λισαβόνα. Είναι απαραίτητο η Κομισιόν να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλεια στη θάλασσα, να αντιμετωπίσει τη θαλασσια ρήπανση. Επομένως, και τα κατημέλη μαζί με την Κομισιόν φυσικά επέχουν ευθύνε στο να εξασφαλίσουν αυτά τα, αυτούς τους στόχους και θα πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα στοιχεία από τα κατημέλη για την εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή οι τέσσερις φορείς είναι κομβική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να πω ότι αν δούμε την κατάσταση με την ΕΝΣΑ υπήρξαν κάποιες διαδικασίες σε σχέση με ε, διαγωνισμούς πλαισίου που καθυστέρησαν ιδιαίτερα και θα ήθελα να πω ότι εγώ θέλω να δώσω την απόλυτη υποστήριξή μου στην κυρία Ινέσα Αγιάλα και υποστηρίζω την ανησυχία της για να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα προπολογισμό στους τέσσερις φορείς και ιδιαίτερα στην ΕΜΣΑ και αυτό βέβαια μπορεί να έρθει σε σύγκρουση στη συγκεκριμένη περίπτωση του να έχει ευρύτερα καθήκοντα η ΕΜΣΑ μέσα στην κρίση, όταν πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα των προσφύγων, της λαθρεμπορίας ανθρωπίνων όντων στη Μεσόγειο κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκταμίευση του προπολογισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι κάπως ανησυχητική το επίπεδο απορρόφησης, αλλά μπορώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ε, γενική αξιοπιστία των ε, λογιστικών στοιχείων για όλες αυτές τις ενέργειες. Αυτά που λέω λοιπόν για την έμψα εφαρμόζονται και για τους άλλους φορείς, μουτάτης μουτάντης. Γι' αυτό η δική μου πρόταση είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την απαλλαγή για τις ε, υπηρεσίες αυτές για το 2014. Ευχαριστώ και ο Πρόεδρος. Η Καρή Παντέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, ε, στο παρελθόν η Επιτροπή Μεταφορών ε, είχε εγκρίνει διάφορες γνωμοδοτήσεις. Είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωση και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για τα σχέδια μεταφορών με κοινοτική συγχρηματοδότηση και για το Ταμείο Συνοχής και για το Περιφερειακό Ταμείο και όχι μόνο για το RTT, τη διευκόλυνση δέντα στην Ευρώπη ή τα τουριστικά προγράμματα κάποιων δημοσιονομικών γραμμών. Τι γίνεται με την ενημέρωση αυτή λοιπόν, ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την ΑΣΑ, την ασφάλεια, Οργανισμό Ασφάλεια για την αεροπορία. Είπαμε ότι έγιναν προσπάθειες για να μειωθεί η σύγκρουση αρμοδιοτήτων και να αποκατασταθεί διαφάνεια. Έγινε όντως αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σαλίνη, εγώ είμαι ο σκιοδησίγητης από την πλευρά του, των σοσιαλιστών και ξέρετε ότι έχουμε παρουσιάσει μία σειρά από τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας σε σχέση με αυτήν την ε, γνωμοδότηση. Αλλά πρέπει να αναφέρω ότι το ελεκτικό ε, συνέδριο για την έκθεσή του στο, για το 2014 έχει μια διαφορετική δομή με αυτά που παρουσιάσατε εδώ. Εμείς πιστεύουμε πρέπει να υπάρξει μια ειδική πτυχή για τις μεταφορές και σε ό,τι αφορά τα θέματα απασχόλησης στον τομέα αυτό, παίζει σημαντικό ρόλο ο τομέας των μεταφορών και τα ένα, <clears throat> το 1 δισεκατομμύριο που έχει προσδιοριστεί για το 2016. Αυτά τα χρήματα είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία δίνονται για την έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αναφέρουμε και για τον τομέα της ε, καινοτομίας έχουν διαπιστώσει της έρευνας και της έχουν διαπιστώσει κάποια σφάλματα το ελεκτικό συνέδριο και αυτό αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο συγκεκριμένα 4,5% ήταν το ποσοστό σφαλμάτων ιδίως σε ό,τι αφορά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. και στην περίπτωση <clears throat> της ε, DigiMove στην ετήσια έκθεσή της αναφέρονται οι... δεν αναφέρονται όλες οι δαπάνες για τα θέματα των μεταφορών έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος για την ε, διαδικασία διαγωνισμών αλλά δεν έχουν δοθεί όλα τα κονδύλια. Επομένως δεν πρέπει να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2014. Επίσης έχουμε θέσει μια τροπολογία για μια υποσημείωση και ζητούμε από την Κομισιόν να αλλάξει αυτό το σημείο στην έκθεσή της και τέλος το αγαπημένο μου θέμα το αγαπημένο μου πάντα θέμα είναι ο τουρισμός. Εγώ χαίρομαι που όλο και περισσότερο υπάρχουν περισσότεροι που υποστηρίζουν τα προγράμματα αυτά και υπήρξε μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τα θέματα στα Για τον τροποποιημένο προϋπολογισμό είναι 11 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα οποία δίδονται στον τουρισμό και 6, αυτό είναι υποχρέωσεις και 6 εκατομμύρια πιστώσεις πληρωμών. Αυτά όμως δεν ανταποκρίνονται στον πραγματικό ρόλο του τουρισμού στις οικονομίες των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό συμφωνώ με τον εισηγητή ότι αυτό το ποσό θα πρέπει να αυξηθεί. Επίσης, συμφωνώ για το ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιό να καταρτήσει μια μελέτη για την επίπτωση που θα έχουν αυτά τα κονδύλια για την βελτίωση του τουριστικού τομέα. Εγώ θα ένιωθα πολύ καλύτερα λοιπόν αν οι, οι επιτροπές υποστηρίξουν τα πιλωτικά προγράμματα και τα μετατρέψουν σε τελικά, σε οριστικά προγράμματα. Η Ανιέσκα Κατσμίσκα. Thank you very much. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να καλύψω όλους τους ε, τομείς και τις διαφόρους οργανισμούς. Να σας ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ε, μόνιμη υποστήριξή της. Ε, καταρχήν για το περιθώριο σφάλματος, το ποσοστό σφάλματος στον τομέα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι ένας ευρύς τομέας που δεν καλύπτει μόνο τις μεταφορές και αυτό το ποσοστό σφάλματος είναι αποτέλεσμα του προγράμματος Legacy στο τομέα της έρευνας που έχει πολύ περίπλοκους κανόνες. Ωστόσο η Κομισιόν αναγνωρίζει απόλυτα την ανάγκη να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος οπότε θα συνεχίσουμε να έχουμε πολύ αυστηρούς εξάντες εξάντε ελέγχους, να συνεχίσουμε να δίνουμε οδηγίες στους ε, δικαιούχους ώστε να ε, ε, τους λέμε, ποια, τους λέμε ποια είναι τα πιο κοινά σφάλματα για να είμαστε βέβαιοι ότι θα μειωθεί το, το ποσοστό σφάλματος. Αλλά όπως σας είπα πρόκειται για πολύ περίπλοκα προγράμματα όπως το πρόγραμμα πλαίσιο, στο, 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και αυτό θα είναι εναντίον μα. Τώρα, τους διάφορους οργανισμούς να θα ανατρέξω και τα ερωτήματα σχετικά με αυτούς. Πρώτος, το θέμα της διαφάνειας και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων. Η Κομισιόν πάντοτε θυμίζει στα συμβούλια των αποκεντρωμένων ε, οργανισμών την ανάγκη, και εγώ είμαι μέλο τριών αποκεντρωμένων, ε, συμβουλίων τριών αποκεντρωμένων οργανισμών, να προσέχουν τη σύγκρουση συμφερόντων, να βάζουν τα βιογραφικά και τη δήλωση συμφερόντων στα δίκτυα, στα, στα site του. Θα ξεκολουθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Σε περίπτωση σφάλματος η πολιτική είναι έχει αργήσει, αλλά συζητήθηκε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο για την αίρα, μας συγχωρείτε, ε, θα το συζητήσουμε στην πρώτη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ε, συμβάσεις προσωπικού όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα τόσο από το εσωτερικό ε, έλεγχο, λογιστικό έλεγχο της Κομισιόν αλλά και από το Συμβούλιο το λογιστικό έχουν υπάρξει σφάλματα. Από το 2009 δεν έχει καθιερωθεί νέα διαδικασία και υπάρχουν πολλές πιθανότητες στις νέες προσλήψεις που έγιναν πρόσφατα το δείγμα να δείξει ότι οι έλεγχοι αυτοί απέφεραν καρπούς και λειτουργήσαν. Τώρα, το θέμα της τελέχωσης των οργανισμών. Εδώ η Κομισιόν προσπαθεί να αναγνωρίσει παλαιότερες θεμητές ανάγκες των οργανισμών. Το ΕΡΑ ε, περιμένουμε ακόμα την αύξηση του αριθμού του προσωπικού που προβλέπεται όταν θα εφαρμοστεί το επόμενο πακέτο. Προβλέπεται δηλαδή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων από το 2018 και μετά. Για την ε, ΕΑΖΑ και τη στελέχωσή της, εδώ είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, διότι η ΕΑΖΑ ζήτησε επιπλέον προσωπικό που θα χρηματοδοτηθεί από τα τέλη και αυτό τελικά συμφωνήθηκε στον τριμερή διάλογο του προϋπολογισμού και υπάρχει μάλιστα αύξηση του προσωπικού που προβλέπεται από το 2016 και μετά. Και δεν θα επιβαρύνει το προϋπολογισμό του Ένωσης. Για το Shift to Rail ε, με χαρά σας ανακοινώνω ότι η πρώτη πρόσκληση δημοσιεύθηκε πριν από μια εβδομάδα. Η σύμπραξη είναι λειτουργική, δεν έχει οικονομική αυτονομία. Σημαίνει ότι όλες οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται από την Κομισιόν. Και αυτό διότι η διαδικασία για την πρώτη επιλογή του, του διευθυντή δεν ήταν επιτυχής. Η δεύτερη επιλογή θα ολοκληρωθεί στις αρχές του Ιανουαρίου, θα γίνει συμβούλιο διοικητικό το οποίο θα επιλέξει τον, ε, τον διευθυντή τον, ή τον διοικητή και θα πρέπει να είναι πλέον αυτόνομη οικονομικά, ε, αυτόνομη οικονομικά το shift to rail από Απρίλιο ή Μάιο. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία υπάρχουν καλά προγράμματα, είναι καλό να έχουμε έτοιμα από καλά προγράμματα, αλλά βεβαίω θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως θα χρηματοδοτηθούν είτε μέσω του ΣΕΦ είτε μέσω του ΕΦΣΥ. Αναλόγως που εμπίπτουν καλύτερα ή μέσω των διαστατικών ταμείων. Έχουμε πληροφορίες πάντοτε για τη χρηματοδότηση των project και έχουμε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και σύντομα θα είμαστε σε θέση να δείξουμε όλα τα project που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Μέσα σε αυτά θα είναι και οι μεταφορές και θα περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων μέσα στο 16 και σίγουρα εκεί θα μπορεί κανείς να δει τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται. Παρακαλώ οι συζητητές θα θέλουν να πούνε κάτι σύντομα και μετά θα πρέπει να συνεχίσουμε μονάχα στα α, αγγλικά για τους τριλόγους και η συνάντηση των συντονιστών θα πρέπει να, μετα, μεταφερθεί τον Ιανουάριο γιατί δεν προφθαίνουμε πια. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Έχουμε τις ε, παρατηρήσεις αυτές που άκουσα, οι οποίες ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την ε, δική μου πρόθεση για την γνωμοδότηση αυτή. Μονάχα θέλω να σταματώ στην τελευταία παρατήρηση της Κομισιόν που λέει ναι για την ευελιξία, αλλά θέλουμε όσο δυνατόν περισσότερα προγράμματα και σχέδια να χρηματοδοτηθούν με το ΕΦΣΥ. Συμφωνούμε με αυτό, είναι ορθό, αλλά αυτή τη στιγμή το ΕΦΣΥ μπορεί, ελπίζω να μπορέσει να χρηματοδοτήσει ε, πολλά σχέδια, αλλά υπάρχουν μια ορισμένα είδη σχεδίων που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει, εκεί όπου η απόδοση του κεφαλαίου απαιτεί περισσότερο χρόνο, όπως παραγωγή χάρη, στα θέματα των, <clears throat> των σιδηροδρόμων. Για το Shift to Rally βλέπω με ικανοποίηση ότι από το Μάιο θα έχει οικονομική αυτονομία και νομίζω ότι με τη φάση των ε, τροπολογιών θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλα αυτά που δεν έχουμε καταφέρει να συζητήσουμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και τους ε, συναδέλφους μου για τα ερωτήματα και τις διευκρινήσεις και για το ενδιαφέρον που περιστρέφεται γύρω από το θέμα αυτό. Ε, χαίρομαι για τις πρόοδους που επιτέθηκαν, ακόμα και αν έχουν έρθει με κάποια καθυστέρηση σε σχέση με την θέλησή μας για τους φορείς αυτούς. Όπως είπε ο κύριος Φαντεκάπ, και εμείς είμαστε η ουσιαστικά αρμόδια επιτροπή για τέτοιου είδους γνωμοδοτήσεις και κακώς πήγαινε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτή την αρμοδιότητα στο μέλλον. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Προθεσμία για τις τροπολογίες 5 Ιανουαρίου του 2016 στις 14 η ώρα. Τέρμα η πολυγλωσία. Συνεχίζουμε στα αγγλικά. Ευχαριστώ τη διερμηνείς για τα τρία πρόσθετα λεπτά. Και η συνεδρίαση των συντονιστών, όπως είπα, δεν μπορεί να γίνει τώρα θα γίνει στις 25 ε, Ιανουαρίου, αλλά την έκθεση για τους ε, τριλόγους θα την κάνω και κλεισμένο των θυρών, γι' αυτό σας παρακαλώ να φύγετε και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.